Ο Πρόεδρος, αγαπητές φίλοι, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αρχίσουμε την απογευματινή συνεδρίαση. Ευχαρίστως καλωσορίζω όλους και όλους εσάς Ευρωπαϊκό ή ελληνικό είναι αυτό. Ευχαριστώ λοιπόν ορίζω όλες και όλους τους Ισπανούς φίλους μας που εκπροσωπούν περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς ε, από την Ισπανία Πρώτα θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με την έκβαση της συναντήσεως των συντονιστών του σημερινού πρωινού. Αφού εγκρίθηκε το σχέδιο ημερησίας διατάξεως από τους συντονιστές, το, άρθρο, το, συγγνώμη, το θέμα 32 για την αναφορά 0410 του 2014 αναβλήθηκε για προσεχή συνεδρίαση. Σε ό,τι αφορά εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις αποφασίστηκε ότι ο εισηγητής για τη σχετική έκθεση του 2015 της Επιτροπής Αναφορών θα είναι η κυρία θα, Βαλίνα της Ενωτικής Αριστεράς και τη συγχαίρω για την ανάληψη του ρόλου αυτού συστάσεις, οι συστάσεις της Πρόεδρου έγιναν δεκτές με την εξαίρεση τη σύσταση για την ε, αναφορά 1372 του 15 όπου το αίτημα της κυρίας Άουκεν καθώς και 1176 του 15 όπου εγκρίθηκε εκεί το αίτημα της κυρίας Βίσερα. Για την 13-15 του 15 εγκρίθηκε συμβιβασμός. Για θέματα Β από την λίστα Β εξαιρέθηκαν το 1199 του 2015 η 0587, άδεια από το 2014 η 0108 του 15 οι εξή αναφορές θα κλείσουν μετά από την δράση που έχει, αναλυθεί από την, που έχει προταθεί από την κυρία Άουκεν 0539 του 13 2370 του 14 0171 του 15 και 0312 του 2015 επίσης. Σε ό,τι αφορά το εργαστήρι για τις αναπηρίες, συμφώνησε οι συντονιστές να οργανωθεί εργαστήρι για τις αναπηρίες το Νοέμβριο φέτος με τη συνεργασία του Policy Department. Σε ό,τι αφορά δημόσιες ακροάσεις, οι συντονιστές ενέκριναν το χρονοδιάγραμμα των ακροάσεων για τη διαφάνεια στις 31 Ιουνίου φέτος Εκεί θα ε, προσκληθεί και ο κύριος Εμίλιο Δικαπιτάνη ως αγορητής για την ακρόαση σχετικά με εμπόδια στην ελευθερία διακίνησης και ε, εργασίας στην ενιαία αγορά, οι συντονιστές εκλήθησαν να υποβάλουν προτάσεις σχετικά με θέματα και ομιλητές μέχρι τέλη Ιουνίου. από την ομάδα εργασίας ΑΦΚΟ, έκθεση για τον κανονισμό. Η πρόεδρος ενημέρωσε σχετικά με τα απεπραχθέντα της ομάδας εργασίας του το τέλους Μαΐου και ε, από τη συνάντηση με τον κύριο Βίλαντ που είναι πρόεδρος της ομάδας αυτής από την 1η Ιουνίου. Οι συντονιστές συζήτησαν με λεπτομέρειες θέματα όπου δεν σημειώθηκε πλήρη συνένεση δηλαδή σύντομα ψηφίσματα, fact-finding visits και οι κανόνες για την εκλογή του Ombudsman. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία θέση για τα θέματα αυτά και θα ενημερωθεί σχετικά η ομάδα εργασίας της Επιτροπής Συνταγματικών ΑΦΚΟ. Σε ό,τι αφορά μη έγγραφα που έχουν ζητηθεί από την νομική υπηρεσία, σημείωσαν οι συντονιστές τα μη έγγραφα τις ε, υπηρεσίας αναφορών για το παραδεκτό της νομικής υπηρεσίας μάλλον για, την, ε, για το παραδεκτό των αναφορών το επόμενο θέμα ήταν ε, επίσκεψη στη Σλοβακία για εξέταση θεμάτων εγκρίθηκε το πρόγραμμα και η σύνθεση έξι επίσημα μέλη και έξι ανεπίσημα και για το δίκτυο της Επιτροπής Αναφορών σημείωσαν συντονιστές τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου και εκλήθησαν να υποβάλουν και άλλες συστάσεις, εάν αυτό είναι απαραίτητο, μέχρι τις 9 Ιουνίου. Η έκθεση από την ομάδα εργασίας για την ευημερία των παιδιών. Αυτό αναβλήθηκε. Αυτά νομίζω ήταν όλα. Αυτά ήταν ε, ε, του σημερινού πρωινού. Μια πραγματικά πολύ χρήσιμη συζήτηση που διεξήχθη μεταξύ μας. Θα ήθελα τώρα να προχωρήσουμε με τη συζήτησή μας. Αν μου επιτρέπετε θα επανέλθω στην πρώτη μου γλώσσα που είναι η Ουγγρική. Πριν να το κάνω αυτό θα παρακαλέσω τους εκπροσώπους των αναφερομένων για την αναφορά 73508, Καστανιέρη και άλλους, που έχουν συλλέξει έναν αριθμό υπογραφών για την συνδρομική σύνδεση, καθώς και την αναφορά 72611 του Ενρίκο Βενέζια για την δημιουργία συνδρομικής συνδέσεως μεγάλης ταχύτητας και 10-26-14 Μάρκο Μπάλα Ιταλού για την ανατροπή της αποφάσεως για την κατασκευή της ταχειας ιδεοδρομικής σιδηροδρομικής συνδέσεως Μιλάνου-Τουρίνου. Ε, καλώς ήρθατε, εσείς αναφερόμενοι, σας δίνω τον λόγο, θα σας παρακαλέσω πρώτα να ομιλήσετε βεβαίως όχι περισσότερα από 5 λεπτά. Ορίστε, έχετε τον λόγο. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Μάρκο Μπάβα και σήμερα εδώ μιλώ εκπρόσωπος ε, της ε, Ένωσης Νέο Μοντέλο ανάπτυξης, τελεία είτε, nuovo μοντέλο τη Βιλούπο, είτε. Για να ζητήσω να ελέγξετε την ε, ε, γραμμή υψηλή ταχύτητα. Ε, Ιταλοί και Γάλλοι πολίτε έχουμε ενωθεί σε αυτή την ένωση για να ζητήσουμε να ελέγξετε τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ που σήμερα έχουν δεσμευθεί για ένα νέο οριστικό project το οποίο περιορίζεται αποκλειστικά στο βασικό, στη βασική σύραγγα και τη τελική του έξοδο μέχρι το Μπουσολένο. Μέσα στην Ιταλική επικράτεια πρόκειται μόνο για 18 χιλιόμετρα, ενώ για το υπόλοιπο της γραμμής ε, γίνεται αναφορά σε μια γενική μελλοντική προσαρμογή της υπάρχουσας σιδηροδρομικής γραμμής. Το 2014 στο Φρέγιους, ε, πέρασαν 3 εκατομμύρια 3 δισεκατομμύρια ε, τόνοι ε, εμπορεύματα για να δικαιολογηθεί το έργο στην ανάλυση κόστος ωφέλους της νέας γραμμής των Ρινολιών. Ε, λένε ότι εντός 7 ετών θα πρέπει να περάσουν 19 εκατομμύρια τόνοι εμπορεύματα αύξηση δηλαδή διαστημικών διαστάσεων, εγώ θα έλεγα πως είναι αδύνατον, της τάξης του 479% σε σχέση με το 2000. 2014 εκτός κάθε πραγματικότητας. Σε μια σύγκριση ανάμεσα σε ένα εμπορικό τρένο που χρησιμοποιεί τη νέα γραμμή και ένα που χρησιμοποιεί την ιστορική πάρουσα γραμμή, το κόστος της ενέργεια της νέας δομής είναι τεράστιο και απαιτεί μια κίνηση, μια ροή που καμία ανεξάρτητη μελέτη δεν θεωρεί να, πιθανό να υλοποιηθεί στις επόμενες δεκαετίες. Μόνο στα πρώτα 400 μέτρα βασικής εξκαφής στην Ιταλική επικράτεια προβλέφθηκαν 160.000 κυβικά μέτρα υλικού που περιέχει αμίαντο. Έτσι λέει στο οριστικό σχέδιο ο διαγωνισμός για το η η οποία θα είναι σύραγγα εξυπηρέτησης στο Πιεμόντε, που μέχρι στιγμής έχει σκαφεί κατά το ίμιση, έχει ανατεθεί στην, στον όμιλο CMC από τη Ραβένα, που κατασκευάζει σε ολόκληρο τον κόσμο κάθε είδος υποδομή και δεν θα έχει πρόβλημα τη στιγμή που στη θέση της τρύπα για το τρένο ψηλής ταχύτητας θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει ε, το ίδιο ε, συγκεκριμένο κόστος με, για, αιωλικές, ε, για μήλους, για συγκεκριμένες πλατφόρμες άφηξης, για φωτοβολταϊκά κόστη με ενέργειας μηδενικά. Από τις αρχές του χρόνου έχουν έρθει στην Ιταλία 46.000 πρόσφυγες, μόνο 15.000 την τελευταία εβδομάδα και προβλέπουμε πως μέχρι τα τέλη του χρόνου θα είναι περίπου 500.000 και αυτό θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι την εισήγηση αυτής της πολιτικής της παραγωγής που σημαίνει ενέργεια και εργασία. Θα δώσει δηλαδή ε, πόρους στην ενέργεια την ανανεώσιμη με τα πολεμικά πολλοί Ιταλοί έχουν ε, μεταναστεύσει στις Ηνωμένε Πολιτείες της Αμερικής. Ε, χρησιμοποιούνται τα χρήματα αυτής της ε, γραμμής τρένου υψηλή ταχύτητας για το Τωρίνο Λιόν, 8 δισεκατομμύρια ευρώ για άλλους σκοπούς. Τα κονδύλια αυτά χρησιμοποιούνται για αυτές τις πλατφόρμες που σας είπα, ε, και θα πρέπει να, ε, για να ολοκληρωθεί ο υγειονομικός και διοικητικός έλεγχος των προσφύγων πριν να μπουν στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Κύριε Γκούντερ Έρτλ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχετε το λόγο. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Λέγομαι Άτλ στη Γενική Διεύθυνση Mobility and Transport της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λαμβάνω το λόγο για να απαντήσω στην πρώτη αναφορά της ημερήσιας διάταξης για, το νέο, για την ε, συνδεση σύνδεση Λιών-Τουρίνο. Αν κατανόησα καλά, ο αναφερόμενος αναφέρει τρία σημεία. Τον όγκο των μεταφερομένων εμπορευμάτων στην ιστορική σιδηροδρομική γραμμή που κατά τη γνώμη του δεν δικαιολογεί τη δημιουργία νέας σιδηροδρομικής γραμμής. Υπάρχουν μεγάλες ποσότητες αμοιάντου και θεωρεί ότι τα χρήματα μπορούν να τοποθετηθούν καλύτερα. Δηλώνω Πρώτα, ότι όλα τα μεγάλα έργα υποδομής στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτελούνται από τις χώρες μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρχίσει ακόμη να ασχολείται με κατασκευή έργων υποδομής. Πρόκειται λοιπόν για έργο το οποίο έχουν αναλάβει να κατασκευάσουν Γαλλία και Ιταλία από κοινού. Το έργο λαμβάνει συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2007 έως 2013 και πιθανώς θα λάβει συγχρηματοδότηση και για την περίοδο 2014 έως 20. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν και εν προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουν άμεση δυνατότητα επιρροής για το εάν θα κατασκευαστεί το έργο ή όχι. Τούτου λεχθέντος βέβαια υπάρχουν αυστηρές συνθήκες αυτοί, όροι για την λήψη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ αυτών και ότι το έργο πρέπει να έχει θετική ανάλυση κόστους κόστους-οφέλους να έχει περάσει όλες τις εθνικές διαδικασίες. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν και περιβαλλοντικές μελέτες και όλα αυτά τα οποία πρέπει να είναι θετικά. Το έργο πρόσφατα απετέλεσε αντικείμενο και στην διάσκεψη κορυφής του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Ολάντ και του Ιταλού Πρωθυπουργού Ρέντσι, οι οποίοι συμφώνησαν να συνεχίσουν ε, την κατασκευή του έργου αυτού που είναι ζωτική σημασία όχι μόνο για Γαλλία-Ιταλία αλλά και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλω να επισέλθω σε όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες και τα σχετικά επιχειρήματα που προβάλλονται σε διάφορες και ποικίλε συζητήσει. Το φορτίο που μεταφέρεται από μια ιστορική σιδηροδρομική γραμμή δεν μπορεί να είναι επιχείρημα. Η ιστορική γραμμή είναι του 1860. Είναι πολύ ιστορική σιδηροδρομική γραμμή διότι ε, για αυτήν φτιάχτηκε η πρώτη σύραγγα στις Άλπεις. Η πρώτη σύραγγα που κατασκευάστηκε στις ε, Άλπεις 1860 ήταν ένα πραγματικό, ε, ένας πραγματικός άθλος και εξακολουθεί να περνάει από την κοιλάδα Σούσα 150 ε, χρόνια αργότερα. Αν φτιαχτεί ένα τέτοιο έργο θα έχει βεβαίω απήχηση και στα επόμενα 150 χρόνια και τότε θα έχει κάνει σωστά τη δουλειά της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το νέο, η νέα σύραγγα λέγεται flat-based διότι η άνοδος είναι της τάξης του 33 της χιλής και όσοι γνωρίζουν από σιδηροδρόμους γνωρίζουν ότι αυτό είναι μια πολύ ε, απότομη ανωδική πορεία. Δεν μπορούν λοιπόν τα τρένα να περνούν από αυτή τη γραμμή για τη διασύνδεση Λιών Τουρίνου. Η νέα σύραγγα βεβαίως θα προσελκύσει και ε, νέες μεταφορές. Δεν φτιάχνει κανείς ωστόσο νέες υποδομές μεταφορών επειδή κοιτάζει εξώ το παράθυρο και βλέπει μα υπάρχουν τόσα πολλά αυτοκίνητα και τροχοφόρα που περνούν ή να κοιτάξει το παράθυρο και να πει «Α, δεν υπάρχουν πολλά, δεν χρειαζόμαστε νέα σύραγγα». Υπάρχουν, ε, υπάρχει πολύ μεγάλος όγκος μεταφορών που περνάει από την Ελβετία ή από την, ε, από τους Ιταλικούς αυτοκινητοδρόμους που περνούν παρακτίως, που είναι όμως υπερφορτωμένοι. Ενώ σωστό είναι να μεταφερθεί και πάλι στον άξονα Λιών Τουρίνου. Και το να δοθούν τα χρήματα αλλού, να τοποθετηθούν αλλού, αυτό δεν είναι υπόθεση για μένα. Αυτό είναι ένα μέγα θέμα το οποίο αποφασίζουν οι πολιτικές ηγεσίες, το που θα επενδύσουν τα χρήματά τους. Νομίζω θα αρκεστώ σε αυτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Αρχίζει η συζήτηση. Ρωτώ τις και τους συναδέλφους, ποιος επιθυμεί να προσθέσει κάτι. Εσείς. Ευχαριστώ, η κυρία Βάλη. Ευχαριστώ. Πρόκειται για ένα έργο, ένα project που χρονολογείται ε, εδώ και 20 χρόνια. Η Ιταλία και η Γαλλία προσπαθούν να το υλοποιήσουν και συνεχίζουν να ε, το παρουσιάζουν στον Ιταλικό και Γαλλικό λαό ω ένα έργο που είναι απαραίτητο να γίνει γιατί θα φέρει τρομερά και φοβερά ωφέλη στην περιοχή. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου και δεν συμφωνούν και χιλιάδες άλλοι. Ε, άνθρωποι που ζουν σε αυτή την ε, περιοχή τόσο από την Ιταλική όσο και από την Γαλλική πλευρά που έχουν κάθε δικαίωμα να εισακουστούν ε, στα αιτιά τους και στις αιτιολογίες και μέχρι στιγμής δυστυχώς δεν είχαν απο... επαρκώς αυτή τη δυνατότητα. Σήμερα λοιπόν κατά μένα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε αυτές τις αναφορές εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο ε, θεωρώντας πως ο αγώνας κατά αυτού του έργου είναι ένας αγώνας που συνεχίζεται εδώ και πολλά χρόνια και που μάλιστα πρόσφατα έλαβε ιδιαίτερη προσοχή από πλευράς άλλων επιτροπών και ο συνάδελφος Μάρκο ε, Βάλι θα σας τα παρουσιάσει τα όσα έγιναν ε, από οικονομικής άποψης. Εγώ θα ήθελα να σας πω κάποια γενικότερα πράγματα που αφορούν, τη συμμετοχή και τη διαφάνεια όσον αφορά αυτό το project. Καταρχάς, θα ήθελα να ρωτήσω με ποιο τρόπο η Κομισιόν εγγυάται τη σωστή εφαρμογή ορισμένων από τις οδηγίες που έχουμε εδώ ορίσει ε, καταρχάς την οδηγία που αφορά την πρόσβαση του κοινού στις ε, περιβαλλοντικές πληροφορίες, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αυτές οι οδηγίες ε, συμβάλλουν στην εφαρμογή της σύμβασης του άρχους που ορίζει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού και τη συμμετοχή του, ιδιαίτερα όσον αφορά projects τα οποία είναι διασυνοριακά, όπως αυτό. Θα ήθελα μάλιστα να θυμίσω σε όλους ότι αυτό το project είναι ακόμα σε φάση μελέτης. Από τη στιγμή που η σύραγγα που έχει μέχρι στιγμής ε, έχει ε, υλοποιηθεί, είναι ε, μία σύραγγα αρχική. Δεν κατασκευάζεται λοιπόν ακόμα. Έχουμε χρόνο δηλαδή να εξετάσουμε σοβαρά και τίμια ποια μπορεί να είναι τα προβλήματα καθώς και να ακούσουμε τους λόγους για το όχι. Στη διάρκεια των ετών λοιπόν το όχι έχει μπει κατά μέρος ε, γιατί στη διάρκεια αυτών των ετών το παρατηρητήριο της κοιλάδα Σούζα που δημιουργήθηκε από το 2006 ως ένας χώρος η αντιπαράθεση συζήτησης για αυτή την επικράτεια στο να μπορέσουν να αναλυθούν ε, τα πλονεκτήματα αλλά και ο κοινωνικός και επιβαλλοντικός αντίκτυπος αυτού του έργου με βίαιο τρόπο ε, ε, κατά κάποιο τρόπο αναγκάστηκε να σιωπήσει γιατί οι εκπρόσωποι του αποκλείστηκαν. Πρόκειται για Δήμου της ίδια αυτή τη Κοιλάδα. Έχουμε 43 δήμους που αντιπροσωπεύουν πάνω από 100.000 κατοίκου, 100.000 κόσμος ζει σε αυτή την περιοχή και στη διάρκεια όλων αυτών των ετών δεν μπόρεσαν να εκφράσουν τη γνώμη τους κατά αυτού του έργου που είναι ένα έργο που επιβάλλεται εκ των άνω από, τις από την κυβέρνηση τη Ιταλία και μέσω τη στρατιωτικοποίηση τη περιοχή η κοιλάδα Σούζα, ακόμα και η περιοχή της εκμετάλλευσης της Σύρακας είναι στρατιωτικοποιημένη με πάνω από 2.000 ε, στρατιωτικούς αστυνομικούς που παρακολουθούν και ελέγχουν την ε, ε, περιοχή. Και θεωρείται και μάλιστα ορίστηκε ως περιοχή εθνικής στρατηγικής σημασίας με ένα διάταγμα του 2013. Και δεν σταματά εδώ η υπόθεση. Υπάρχουν ένα σωρό άλλα στοιχεία που δείχνουν ότι δεν πρόκειται για ανοιχτή και τίμια ε, διαβούλευση με το κοινό. Ο πρώην πρόεδρος μάλιστα αυτού του παρατηρητηρίου της Βάλντε Σούζα ε, είναι υποδικαστική δικαστική δίωξη ακριβώ επειδή δεν έδωσε πρόσβαση στις πληροφορίες ε, για, σε αυτούς τους Δήμους που είναι κατά της υλοποίηση του έργου. Οι δικαστικές διαδικασίε θα συνεχιστούν, θα ακολουθήσουν την πορεία τους. Έχουμε και αυτό τον λόγο για να διατηρήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις της υπόθεσης αυτής. Και θα ολοκληρώσω αναφερόμενοι στα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ή στην υποτιθέμενη αυτή ανάγκη να πληρωθεί αυτή η ελλειπής σύνδεση. Λες και δεν υπάρχει ε, σιδηροδρομική γραμμή που να λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Και σήμερα μάλιστα υπολειτουργεί. Λέτε για κορεσμό της γραμμής, πόρο απέχουμε από το κορεσμό της γραμμής που συνδέει το Τωρίνο με τη Λιόν. Και τέλος θα ήθελα να σημειώσω στους συναδέλφους για τη λέγεται ότι η μεγάλη ταχύτητα χρησιμοποιείται σε ολόκληρο τον κόσμο για τους επιβάτες. Σκεφτείτε ας πούμε τη σύνδεση ανάμεσα στο Τωρίνο και τη Λιόν που σήμερα μεταφέρει γύρω στις 2.000 ε, ε, ανθρώπους ημερησίως. Είναι πολύ μικρά νούμερα όταν μιλάμε για άλλα μέρη του κόσμου που έχουμε 40.000 επιβάτες την ημέρα που μεταφέρονται. Και το μέγα ψέμα αφορά ακριβώς τη χρήση της υψηλής ταχύτητας για τα εμπορεύματα, για φορτία. Είναι τρέλα αυτό το πράγμα. Ότι θα χρησιμοποιηθούν τα τρένα υψηλής ταχύτητας για τα... τη μεταφορά φορτίων. Και οι προβλέψεις για το μέλλον λοιπόν δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, γιατί ακριβώς τα τελευταία 16 χρόνια είδαμε δραστική μείωση των ε, εμπορικών ε, μεταφορών ε, μέσω σιδηροδρόμων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε τόσο μεγάλα project να μπορούμε να αξιολογούμε με ξεκάθαρο και ανεξάρτητο τρόπο ποια είναι τα ωφέλη που μπορεί να αποφέρει μια υποδομή σε μια περιοχή ε, χρησιμοποιώντας αυτό που λέγεται life cycle assessment, δηλαδή εκτίμηση του κύκλου ζωής ενός έργου και το ωφέλη που μπορεί να αποφέρει σε μια περιοχή. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, είναι απαραίτητο να γίνει, ωστόσο εγώ ζητώ και κάνω και μια πρόταση προφανώς να παραμείνει ανοιχτή αυτή η ε, αναφορά, να μπορέσουμε να στείλουμε μια επιστολή στις Ιταλικές και Γαλλικές αρχές, ώστε να θίξουμε τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι διάφορες αναφορές και επιπλέον εγώ προτείνω και μια επίσκεψη σε αυτήν την περιοχή, σε αυτό το εργοτάξιο, τόσο από την Ιταλική πλευρά όσο και από την Γαλλική, για να ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους που εδώ και 25 χρόνια αγωνίζονται κατά αυτού του έργου. Διότι δεν είναι δυνατόν τα δικά τους ε, προβλήματα να μην έχουν εισακουστεί εδώ και τόσα χρόνια. Ευχαριστώ. πολύ, κυρία μου. Μάλιστα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν είναι πρώτη φορά που συζητάμε στο Κοινοβούλιο για αυτά τα έργα, γιατί είναι και ένα από τα πιο δαπανηρά ε, έργα που χρηματοδοτεί ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν μέρη. Ε, γι' αυτό και στηρίζουμε εντόνως την αναφορά που φθάνει από την Ιταλία και επικρίνουμε εντόνως το project για τέσσερις βασικούς λόγους. Πρώτον, δεν είναι δημοκρατικό, δεν είναι διαφανές, είναι άχρηστο και επικίνδυνο. Και θα εξηγήσω γιατί δεν είναι δημοκρατικό, γιατί όπως ξε... σας εξήγησε η συνάδελφος Λεωνόρα Εύη, υπάρχουν ε, ε, συγκεκριμένοι δήμοι που είναι εντόνως ε, κατά και δεν έχουν ποτέ ακουστεί. Είναι ένα είδος δικτατορικού καθεστώτος προς... για την εφαρμογή ενός project χωρίς να δοθεί καμία σημασία στον κόσμο που ζει εκεί και που θέλει να δώσει τη γνώμη του για το συγκεκριμένο έργο. Δεν είναι διαφανή η κατάσταση, γιατί δεν υπάρχουν ανεξάρτητε εκτιμήσει και συγκεκριμένε πιστοποίησει για το κόστο. Έχουμε ένα έργο δισεκατομμυρίων, αλλά οι αξιολογήσει έχουν γίνει από μη ανεξάρτητου οργανισμού, από εταιρείε που μετά Βλέπουμε ότι εντάσσονται σε σύγκρουση συμφερόντων, ανθρώπους που διαχειρίζονται την ε, εταιρεία που κάνει την αξιολόγηση και την εταιρεία που υλοποιεί το έργο. Ε, άρα λοιπόν δεν υπάρχουν ε, ανεξάρτητες αξιολογήσεις για αυτό το έργο. Θέλουμε δηλαδή να χρηματοδοτήσουμε ένα έργο και μετά θα βρούμε και ένα τρένο που δεν θα μεταφέρει ούτε φορτία ούτε επιβάτες. Θα έχουμε δηλαδή δαπανήσει ένα σωρό χρήματα για ένα άχρηστο έργο το οποίο θα έχει δημιουργήσει και προβλήματα στην περιοχή που δεν το θέλει. Δεν είναι διαφανές το έργο γιατί δεν, έχουν υπάρχει, δεν υπάρχει καμία διευκρίνηση. Εγώ είμαι συντονιστή στην ομάδα μου, ζητήσαμε ε, πληροφορίες για τις διάφορους διαγωνισμούς, ε, τις διάφορους μειοδοτικούς διαγωνισμούς, γιατί ένα τέτοιο, για μια τέτοια σύραγγα γίνονται καταρχάς διαγνώσεις. Ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός εν μέρη χρηματοδοτεί το συγκεκριμένο έργο και δεν δίνονται στοιχεία, γιατί τα κράτη-μέλη, Γαλλία και Ιταλία, το θεωρούν δικό τους. Επειδή όμως το Ευρωκοινοβούλιο είναι 28 κράτη και τα χρήματα για τη χρηματοδότηση του έργου είναι και των 28. Η Επιτροπή Προϋπολογισμού ζήτησε αυτά τα αρχικά έργα και τις αρχικές διαγνωστικές εργασίες και με μεγάλη ε, ε, ε, πλειοψηφία για το 2014 ζητήσαμε πλήρη διαφάνεια για τις οικονομικές πληροφορίες για το τρένο ψηλής ταχύτητας το Ρήνο Λιών. Δεν έχουμε ακόμα τις πληροφορίες, είμαστε σε στενή επαφή με τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ την αρμόδια για να πάρουμε αυτές τις πληροφορίες. Έπειτα είναι άσκοπο και άχρηστο γιατί δεν υπάρχουν αρκετές μεταφορές φορτίων που να αιτιολογούν ένα τέτοιο έργο και έπειτα ε, στα προκαταρκτικά έργα ήδη ε, υπάρχουν ε, δικαστικές διαδικασίες για απάτη αλλά και για διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος, ε, της μαφίας. Πολύ επικίνδυνο να ξεκινήσει τόσο τεράστιο έργο όταν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις και ειδικά όταν πρόκειται για διασυνοριακό έργο υπάρχουν διαφορές δικαίου ανάμεσα στη Γαλλία και στην Ιταλία και δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς ποιο είδος δίκαιο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και ανού κράτου δίκαιο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα. Όπω καταλαβαίνετε, το οργανωμένο έγκλημα εκεί θριαμβεύει. Πώ θα χρηματοδοτήσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το οργανωμένο έγκλημα με αυτόν τον τρόπο. Για αυτού του λόγου λοιπόν εκφράζουμε τη λύπη μα για αυτό το έργο και θα θέλαμε αυτή η αναφορά να μείνει ανοιχτή και να αναλυφθούν πρωτοβουλίε από το Ευρωκοινοβούλιο για να χυθεί φως σε αυτή την υπόθεση και όλοι στην Ευρώπη να καταλάβουν πόσο άχρηστο είναι αυτό το έργο και πόσα άλλα μεγάλα έργα είναι άχρηστα, πού θέλουμε να υπάρξει διαφάνεια. Δεν θέλουμε πια ε, τρένα χωρίς επιβάτες ή φορτία, αυτοκινητοδρόμους ε, άδειους από αυτοκίνητα. Δεν θέλουμε πια τέτοιου είδους σπατάλες, ούτε και προβλήματα με τη δημοκρατία, γιατί εδώ επιβάλλεται ένα έργο σε μια ολόκληρη περιφέρεια του Πιεμόντε, που είναι η Βαλ Σούζα. Ο κύριος Πέτερ του Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ. Το γενικό πρόβλημα είναι ότι βεβαίως δεν υπάρχουν μεγάλα έργα που να μην αντιμετωπίζουν κριτική. Μέχρι τώρα η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και κατανοητή. Δηλαδή έχουμε πει θέλουμε μεγάλους, μεγάλους άξονες μεταφορών μεταξύ νότου, βορρά κτλ. Αλλά όλα αυτά τα κάνουμε σε στενή συνεργασία με τις χώρες μέλη, διότι αυτές τελικώς θα εκτελέσουν τα έργα. Αυτό σημαίνει βέβαια επίσης ότι οι χώρες μέλη διεξάγουν τον διάλογο με τους πολίτες. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή. Δεν υπάρχει κανένα μεγάλο έργο το οποίο να μην αντιμετωπίζει κριτική και βεβαίως έχει παρεμπίπτου σε συνέπειες η κατασκευή του κτλ. Τώρα θα ήθελα να επανέλθω στα επιχειρήματα των προσώπων που ήδη μίλησαν αλλά θέτω και το ερώτημα πώς θα λύσουμε το πρόβλημα. Πρώτα-πρώτα είναι χρήσιμο το έργο. Ομολογώ ότι δεν είμαι σε θέση να το κρίνω από εδώ, εάν δηλαδή οικονομικός είναι αναγκαίο. Εδώ νομίζω πρέπει να διευκρινιστεί στον διάλογο μεταξύ των δύο χωρών μελών, Γαλλίας-Ιταλίας. Αν χρειάζονται και άλλες πληροφορίες εκεί, εκεί έστω να το εξετάσουμε. Τώρα, αν κάποια πράγματα σημειώθηκαν σφάλματα, δηλαδή στην ε, προκήρυξη του έργου, αυτό πρέπει να το κρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βεβαίως αν υπάρχει υπόνοια διαφθοράς. Η ερώτηση που θέτω τώρα είναι πώς θα λύσουμε το πρόβλημα χωρίς να παίξουμε πινκ-πονγκ. Εγώ θεωρώ ότι ένα μέρος του προβληματισμού πρέπει να λυθεί και από τις τοπικές αρχές. Δεν ξέρω εάν υπάρχουν και στην Ιταλική και στην ε, Γαλλική Βουλή Επιτροπή Αναφορών και βεβαίω και συνήγοροι του πολίτου που να ασχοληθούν. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα για τα οποία εμείς είμαστε αρμόδιοι και να δούμε για ποια είμαστε αρμόδιοι και για ποια δεν είμαστε και που πρέπει δηλαδή να αποταθούμε για την εξέταση σε άλλους. Ξαναλέω ότι βεβαίως τα μεγάλα έργα υποδομών έχουν σημαντικές συνέπειες και βεβαίως αντιμετωπίζουν κριτική. Και κυρίως ο διάλογος με, τις, με τους τοπικούς παράγοντες είναι σημαντικός. Καταλαβαίνω και αυτό που αντιτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι καταρχήν αρμόδιες είναι οι χώρες μέλη και αυτές ε, φέρουν τη βασική ευθύνη. Αρκούμε σε αυτά εισαγωγικώς, δηλαδή ως αρχική παρατήρηση, και ε, να δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στους αναφερόμενους. Ευχαριστώ. Κύριε Βαλίνα. Ευχαριστώ και εγώ. Καλησπέρα. Και εμείς από την ΚΟΕ στηρίζουμε την αναφορά αυτή. Γιατί από ό,τι φαίνεται τα πράγματα και τα νούμερα δεν είναι πολύ ξεκάθαρα. Μας έχουν φέρει σύντροφε από την Ιταλία νούμερα που λένε ότι από το 2011 έχει αυξηθεί πάρα πολύ η κυκλοφορία. Το 83, 9,8 εκατομμύρια τόνοι. Ενώ το 2014 ήταν 13,2 εκατομμύρια. Επίσης είναι αυτή η διαδρομή, είναι 57 χιλιόμετρα παραπάνω. Ήδη το 2012 το δικαστήριο της Γαλλίας είπε ότι η γραμμή αυτή θα έπρεπε να περιοριστεί, να μειωθεί η κυκλοφορία. Όμως το τούνελ αυτό έχει ακόμα δυνατότητες, αλλά αν υπάρχει κρίση τότε καλά θα κάνουμε τα χρήματα να τα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα. 15 με 17 εκατομμύρια τόνοι Κυκλοφορούν λοιπόν ανάμεσα στην Ελβετία και την Αυστρία χωρίς πρόβλημα λένε μέχρι τώρα. Στην Ισπανία έχουμε αρκετή εμπειρία με αεροδρόμια χωρίς αεροπλάνα, με ε, αυτοκινητοδρόμους οι οποίοι μένουν άδειοι γιατί έχουν φτιαχτεί χωρίς να χρησιμεύουν σε τίποτα. Οπότε πρέπει να καταδείξουμε ότι τελείωσε πια αυτή η περίοδος της πατάλης και των άχρηστων έργων. Άρα την αναφορά αυτή πρέπει να την αφήσουμε ανοιχτή, αλλά και επιπλέον να δώσουμε την αναφορά αυτή και στην ΕΝΒΗ και στην ΤΡΑΝ και σε αυτές τις κοινοβουλευτικές επιτροπές μεταφορών και περιβάλλοντος. 40% των χρημάτων των Ευρωπαίων, Ιταλών, Γάλλων και των υπόλοιπων χωρών ε, σπαταλώνται. Νομίζω ότι αυτή η νοοτροπία των μεγάλων έργων που δεν αποδεικνύεται η αναγκαιότητά τους, όπως πολύ καλά το έλεγαν και οι συνάδελφοι, μετά το θα γίνει και με τα τρένα και με τα αεροπλάνα. Ε, αυτή η κουλτούρα λοιπόν, αυτή η νοοτροπία φτάνει πια χωρίς έλεγο. Και να ξέρουμε, είναι αναγκαία τα έργα. Α, ναι, έχει καλώς και επίση να λάβουμε υπόψη μα και τον αντίκτυπό τους, ο οποίος έτσι κι αλλιώ ε, δεν έχει επιστροφή. Ο Μαρία. Μαριάς. Κύριε Πρόεδρε, ακούσαμε με ενδιαφέρον τους ε, αναφέροντες και φυσικά τους συναδέλφους ε, από την Ιταλία, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα το θέμα. Εγώ αυτό που έχω δει και παρακολουθώ αρκετά χρόνια είναι ότι υπάρχουν πάντοτε αντιδράσεις ε, γύρω από την λειτουργία αυτής της ε, συγκεκριμένης ε, σιδηροδρομικής γραμμής. Και κυρίως υπάρχουν αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες κάθε φορά παραπονούνται ότι δεν ενημερώνονται, ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η ίδια τους η θέση και ότι οι αρχές είτε της Γαλλίας είτε της Ιταλίας προχωρούν χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τοπικά τι συμβαίνει. Και ακούσαμε ότι υπάρχουν μια σειρά από δήμοι οι οποίοι δεν έχουν κληθεί στη διαβούλευση. Το θέμα μας αφορά πρώτα απ' όλα διότι τα χρήματα, ένα μέρος των κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται για το έργο είναι χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένω, έχουμε αρμοδιότητα να εξετάσουμε το ζήτημα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι τα έργα τα οποία γίνονται, ε, πάντοτε αυτά τα μεγάλα έργα πρέπει να έχουν και ένα στοιχείο διαβούλευσης όπως ε, προβλέπονται και από τη Σύμβαση Άρχους ε, και από άλλες διατάξεις ε, ε, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι προφανές ότι εδώ αυτό δεν έχει τηρηθεί. Το επόμενο θέμα είναι ότι λένε οι συνάδελφοι ότι το έργο αυτό είναι πάρα πολύ ακριβό ή επίσης ότι δεν χρειάζεται. Σε μια φάση περιορισμού των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν πράγματι αυτό το έργο δεν χρειάζεται διότι υπάρχει μια γραμμή η οποία δεν έχει κορεστεί και η οποία εξυπηρετεί, σημαίνει ότι υπάρχουν δυνατότητες να διατεθούν τα κεφάλαια αυτά σε άλλα έργα, ούτω ώστε να έχουμε ενδεχόμενα σιδηρόδρομο υψηλής ταχύτητας σε άλλες περιοχές. Να επισημάνω πολύ απλά ότι όσοι ταξιδεύουμε και είναι περισσότεροι από εδώ, από τις Βρυξέλλες προς το Στρασβούργο και αντίστροφα κάθε φορά που έχουμε την Ολομέλεια στο Στρασβούργο, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει στην ουσία μια γραμμή υψηλή ταχύτητα από τι Βρυξέλλε προ το Στρασβούργο. Και πάμε και περνάνε αρκετέ ώρε. Αν λοιπόν δεν χρειάζεται αυτή η γραμμή, είναι προφανέ ότι θα μπορούσαν να επενδυθούν τα κεφάλαια αυτά σε άλλε περιοχέ. Υπάρχουν περιοχέ του Νότου, όπω και στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη, που εκεί ίσω είναι πολύ πιο απαραίτητη η επένδυση. Άρα λοιπόν αυτά όλα μας δείχνουν ότι πρώτα απ' όλα εμείς από την πλευρά μας στηρίζουμε την αναφορά. Δεύτερον, επιμένουμε, όπως και οι άλλοι συνάδελφοι, ότι αυτή η αναφορά πρέπει να μείνει ανοιχτή. Το τρίτο είναι ότι σίγουρα πρέπει να ενημερωθούν και άλλες επιτροπές, όπως είναι η ΕΝΒΗ, αλλά ενδεχόμενα και άλλες επιτροπές, budget, ε, του Κοινοβουλίου μας. Και το επόμενο είναι ότι πρέπει να σταλεί επιστολή στην ίδια την Ιταλική κυβέρνηση και την Γαλλική κυβέρνηση, να έχουμε τις αντιδράσεις τους, όπως επίσης φυσικά να σταλούν επιστολές και στους ενδιαφερόμενους δήμους οι οποίοι είναι στην περιοχή και οι οποίοι δεν έχουν κληθεί ε, καθόλου στην όλη διαβούλευση. Επομένως, κλείνοντας, ε, θα έλεγα ότι είναι ένα σοβαρό θέμα, πρέπει να μας απασχολήσει, να μείνει ανοιχτή η αναφορά και να δούμε από εκεί και πέρα, μετά και από αυτές τις προτάσεις που έχω κάνει εγώ και οι συνάδελφοι, πώς θα συνεχίσουμε πάντα στηρίζοντας τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι άλλωστε μας έχουν εκλέξει για να είμαστε εδώ, να στηρίζουμε τις απόψεις τους και τα συμφέροντά τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Πρόεδρε, θέλω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτά που άκουσα από τον κύριο Γιάρ. Είναι αλήθεια ότι κάθε μεγάλη επένδυση πάντα αντιμετωπίζει κριτική. Είναι λοιπόν δύσκολο να πούμε περισσότερο χωρίς να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία για το κατά πόσο επένδυση αυτή είναι αναγκαία ή όχι. Το ξέρω πολύ καλά, γιατί και η Πολωνία σήμερα είναι ένα τεράστιο εργοτάξιο και θυμάμαι πολύ καλά ότι πριν από λίγο καιρό έγινε μια τεράστια επένδυση ε, καλή γενικά μιλώντας, αλλά πέρασε από πολύ σκληρή κριτική. Έχουμε τώρα για το συγκεκριμένο έργο την απάντηση της Επιτροπής του 2012, πριν από τέσσερα χρόνια δηλαδή. Και επιπλέον η απάντηση αυτή του 2012 βασίζεται σε δεδομένα του 2011. Οπότε δεν είμαι σε θέση τώρα να πω κατά πόσο πρέπει να κλείσουμε να αφήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά. Αυτό όμως που πιστεύω είναι ότι πρέπει να έχουμε πιο πρόσφατες πληροφορίες σημερινές για το τι συμβαίνει ακριβώς επί τόπου. Πρέπει δηλαδή να ξέρουμε καταρχήν κατά πόσο όλα γίνονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Γιατί μπορεί εδώ και όλα αυτά τα χρόνια να έχουν προχωρήσει τόσο πολύ τα έργα που αν θέλουμε τώρα να τα κυρώσουμε όλα θα ήταν ακόμα χειρότερη σπατάλη. Δεύτερον, τα χρήματα δαπανώνται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ή έχουν υπάρξει καθυστερήσεις στις πληρωμές. Τρίτον, βλέπω ότι το σχέδιο έπρεπε να τροποποιηθεί, ότι έπρεπε να μειωθεί σε ένα βαθμό. Τι επιπτώσεις ε, έχει αλλαγή αυτή στο κόστος. Και τέλος, όσον αφορά τα γραφειοκρατικά, προκειμένου να υλοποιηθεί η επένδυση αυτή. Όλα αυτά τα τυπικά τα γραφειοκρατικά έχουν γίνει. Και το τελευταίο, Ίσως πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει σημερινές πληροφορίες όσον αφορά την πρόοδο του έργου σήμερα. Μετά από 3,5 χρόνια από τότε που έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί τα έργα. Οι πληροφορίες αυτές είναι ζωτικής σημασίας. Αν έχει προχωρήσει πολύ το έργο δεν πρέπει να το σταματήσουμε γιατί τότε θα ήταν χειρότερη σπατάλη αυτή. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανέναν άλλον επιθυμεί να λάβει το λόγο ε, εκ των συναδέλφων. Εκ των συναδέλφων, κύριε Μπάβα, εσείς. Να απαντήσω αμέσω ε, σε τελευταία αυτή τη συζήτηση. Όπως είπα ήδη, τα έργα βρίσκονται στην αρχή. Έχουν ίσα ίσα ξεκινήσει. Οικονομική ε, εξηγήσει. Και εδώ απαντώ αμέσως και τον εκπρόσωπο της Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Σας καλώ να δείτε ότι αν δεν υπήρχαν οι χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανέρχονται ήδη σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ, ούτε η Ιταλία ούτε η Γαλλία θα είχαν βάλει φράγκο. Ε, Υπάρχει ρητή βούληση, τουλάχιστον όσον αφορά την Ιταλία, γιατί η Γαλλία δεν μπορώ να πω, αλλά πιστεύω πως είναι το ίδιο, να προσελκύσουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στην επικρατειά τους. Πέρα από το οικονομικό σφάλμα, του να προβλεφθούν οι λύσεις ε, λόγω υποτιθέμενων αναγκών. Άκουσα ότι υπάρχει μία πρόταση και ελπίζω ε, να γίνει η επίσκεψη επιτόπου και να έρθει και ο Υπουργό Μεταφορών. Να δούμε λοιπόν ποια είναι η πραγματική κυκλοφορία και το τι μπορεί να διευθυνθεί στην υφιστάμενη γραμμή. Δεν υπάρχει καμία απολύτω ανάγκη για αυτή τη σύραγγα σε εκείνη την περιοχή. Και να προσθέσω το μόνιμο δικαστήριο των λαών έχει καταδικάσει αυτή, ε, αυτό το έργο. Η Δήμοι είναι κατά, η, ο κόσμος που ζει στην περιφέρεια, στην Ιταλία και στη Γαλλία είναι κατά. Ο μόνος πραγματικός λόγος που εγώ βλέπω και γι' αυτό ακριβώς και καλό την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποσύρει τα κονδύλια είναι ότι υπάρχει υψηλή συγκέντρωση κονδυλίων για άσκοπα και εξαιρετικά δαπανηρά έργα σε μια ζώνη όπου υπάρχει υψηλή συγκέντρωση μαφιών Άρα λοιπόν δεν αποκλείεται καθόλου τα χρήματα της γραμμής ψηλής ταχύτητας να δοθούν όχι άμεσα αλλά έμεσα σε εταιρείε που έχουν, ε, όπου έχει διεισδύσει η μαφία και μέσω από αυτές η μαφία να κάνει ωραιότατα τη δουλειά της σε μια φάση οικονομικής κρίσης που τα κέρδη της φτάνουν, που μάλλον σε αυτή τη φάση κρίσης αγοράζουν διαρκώς εταιρείε για παράνομους σίγουρα σκοπούς Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να ξανασκεφτείτε αυτά τα χρήματα, να τα πάρετε πίσω. Αν πραγματικά αυτά τα έργα εξυπηρετούν το γαλλικό και το ιταλικό κράτος, να τα κάνουν με τα λεφτά της Ιταλίας και της Γαλλίας και νομίζω πως αυτό θα αρκέσει για να σταματήσουν διαπαντός οι εργασίες αυτές και θα σας αποδείξει ότι καμιά από αυτές τις δύο χώρες δεν έχει συμφέρον να κάνει αυτά τα έργα πέρα από μια καθαρά οικονομική επιχείρηση. Ελπίζω πως θα έρθετε επί τόπου και θα μπορείτε να δείτε με τα ίδια σας τα μάτια, θα ακούσετε τους δημάρχους, της Ιταλούς και τους Γάλλους και όπως σας είπα για την Ιταλία είναι όλοι κατά τη υλοποίηση του έργου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, μπορούμε να κλείσουμε το σημείο αυτό ως εξής. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν συνηθίζουμε να λέμε κάτι σε βάρος κάποιου, αλλά τώρα διορθώστε με αν κάνω λάθος αυτά που θα πω. Υπάρχει, από τη μια, μία αναφορά με πολύ σοβαρή κριτική στη συγκεκριμένη περίπτωση για αυτή τη νέα γραμμή, τη σιδηροδρομική το Ρήνο Λιών. Με τις συνέπειες και για το κατά πόσο είναι νόμιμο ή όχι το έργο. Από την άλλη, έχουμε συζητήσει και τι μας λέει η Επιτροπή, ότι πάνε 10 χρόνια. Αν κατάλαβα καλά, πρόκειται για ένα τμήμα της γραμμής Βουδαπέστης-Λιών, για μια νέα σύνδεση σιδηροδρομική ανάμεσα σε αυτές τις δύο πόλεις, άρα δεν πρόκειται για μια επένδυση απομονωμένη, πρόκειται για κάτι που έχει να κάνει με το γενικότερο ευρωπαϊκό δίκτυο, είναι γαλλοευρωπαϊκή υπόθεση. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ίσως να μπορεί να μας πει κάτι και το Συμβούλιο μάλιστα. Γιατί τη γραμμή αυτή που αρχίζει από τη Βουδαπέστη λοιπόν δεν μπορεί να σταματήσει στο Μιλάνο για παράδειγμα αντί να πάει μέχρι τη Λιόν. Οι αναφέροντες μας λένε ότι η σύνδεση αυτή το Ρήνο Λιόν είναι περιττή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πιστεύω ότι μπορεί να απαντήσει πάνω σε αυτό. Και οι δύο κυβερνήσεις, η Ιταλική και η Γαλλική, επίσης μπορούν να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα. Εγώ νομίζω ότι συμφωνούμε λίγο πολύ ότι θα αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά, έτσι. Το δέχεστε όλοι αυτό. Ωραία, αυτό είναι το ένα. Και μετά πρέπει να πάρουμε και άλλη μια απόφαση. Γράψαμε, όπως πρότειναν πολλοί, στις κυβερνήσεις, την Ιταλική και τη Γαλλική, για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις επενδύσεις που έχουν γίνει και ένα άλλο στοιχείο. Η Επιτροπή να μας πει για τη συνέχεια. Έχει νόημα να εκτιμήσουμε τη συγκεκριμένη αυτή επένδυση όταν θα ξέρουμε ακριβώς για τα ποσά. Και το άλλο που είπαν και οι συνάδελφοι είναι να στείλουμε επιστολή και σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές για να συνδεθούν και αυτοί με μας. Παρακαλώ, Πέτερ. Με την έννοια αυτή μπορεί ίσως να διευκρινίσει από την αρχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν όντως υπάρχουν ενδείξεις ότι στη διαδικασία προκηρύξεως του έργου υπάρχουν σφάλματα. Για να είμαστε προστατευμένοι και απέναντι σε οποιασδήποτε ας πούμε εγκληματικές ε, διακλαδώσεις, ας το πω έτσι, του έργου, της χρηματοδοτήσεως του έργου αν δηλαδή οι προκηρύξεις είναι σύμφωνες με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Γιατί οφείλουμε να λάβουμε υπόψη και τις ε, καταγγελίες των αναφερομένων ότι ενδεχομένω υπάρχουν κάποια πράγματα. Άρα, δύο πράγματα. Αναγκαιότητα ημί του έργου. Δεύτερο, θα πρέπει να μην υπάρχει υπόνοια διαφθοράς. Ευχαριστούμε. Ναι. Ε, σωστά και αυτό που λέτε. Ναι. Να συμπεριληφθεί και αυτή η ερώτηση στην επιστολή, στην Επιτροπή. Ωραία. Τελειώνουμε με αυτό το σημείο και περνάμε στο σημείο 11 που είναι η αναφορά dietmann Dietmann-Koll. Σχετικά με τον έλεγχο προπολογισμών, νομίζω ότι Κάτι είχαμε πει γι' αυτό. Ναι. Πράγματι, θα το συνδέσουμε με την Επιτροπή Προπολογισμών. Λοιπόν, το προηγούμενο δηλαδή σημείο. Τώρα πάμε στο σημείο 11. Αναφορά λοιπόν 0974 το 2014 του Dietmar Gold, Αυστριακής Ιθαγένειας. σχετικά με σχεδιαζόμενη συνδρομική γραμμή στο Σάλτσμπουργκ και πιθανέ παραβιάσεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριο Δίτμαρ Γκολτ θα πάρει πρώτα το λόγο για να μας παρουσιάσει την αναφορά του. Λέγομαι Γκόλτ, σα ομιλώ ω εκπρόσωπο της Υπερκομματικής Επιτροπής Πολιτών με τον τίτλο που βλέπετε στην διαφάνεια. Πρώτο, έλαβα πρόσφατα το πρόγραμμά σας, την ημερήσια διάταξή σας δηλαδή για σήμερα. Ελπίζω, γιατί είναι πολύ ουσιώδες, για την κατασκευή του, του αστικού αυτού σιδηροδρόμου, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη και η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην περιοχή αυτή. Γιατί καταθέσαμε την αναφορά. Βάση των, του προβληματισμού μας ήταν ότι η πολιτική περιβάλλοντος Η προσθέτει του περιβάλλοντο περιλαμβάνεται στη Συνθήκη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 174, παράγραφο 2. Και εκεί επιβάλλεται και η αρχή τη πρόληψη. Και βεβαίω όταν σημειώνονται προβλήματα, τα προβλήματα αυτά οφείλουν να λύνονται σύμφωνα με την αρχή του ο ρηπαίνων πληρώνει. Βλέπετε στην διαφάνειά μου τώρα και τη σχετική οδηγία. Για λόγους χρόνου δεν θα επεκταθώ σε αυτήν. Περί τίνος πρόκειται. Είναι περίπλοκο βεβαίως το θέμα. Πρόκειται για την περιφέρεια του Σάλτσπουργκ, στο, ε, στο κέντρο της οποίας βρίσκεται μια πόλη η οποία χωρίζεται από ένα ποτάμι και τρία βουνά. Αυτό κατακαιρματίζει βεβαίως την αστική δομή και σε ό,τι αφορά τις κατοικίες αλλά και σε ό,τι αφορά τις μεταφορές. Παρόλα αυτά έχουν δημιουργηθεί τέσσερις άξονες για την κίνηση και μέχρι τώρα τις τελευταίες δεκαετίες έχουν δαπανηθεί πολύ περιορισμένοι πόροι για τις εγγύς αστικές συγκοινωνίες. Έτσι λοιπόν κυριαρχεί το ατομικό στοιχείο στις μεταφορές με 44%. Αν εξετάσει όμως κανείς προσεκτικότερα την περιφέρεια, θα ειδεί ότι σε μια κτίνα 50 χιλιόμετρων από το αστικό κέντρο ζουν ένα εκατομμύριο άνθρωποι και αν επεκτείνεται την περιφέρεια αυτή περισσότερο φτάνεται στα 17 εκατομμύρια ανθρώπων, μια περιφέρεια δηλαδή σημαντική. Η επικαιρότητα έχει ως εξής. Φέτος, και θα επανέλθω σε αυτό αργότερα, και ο Δήμος και το κρατήδιο δεν έχουν κάνει σχεδόν τίποτε για τις δημόσιες μεταφορές. Μέχρι το 1953 αυτή ήταν η εικόνα που δίναμε, που δέτε στη φωτογραφία, που δεν είναι πλέον επικαιρή, τώρα στα ε, προβλήματα περιβάλλοντος που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Εμείς έχουμε τονίσει ένα πρόβλημα, δηλαδή τις τιμές οξυδίων του αζότου. Βλέπετε στο γράφημα από το κρατήδιο του Σάλτσπουργκ ότι έχουμε δύο σημεία μετρήσεως όπου περιλαμβάνονται τα οξύδια του αζότου, τα οποία υπερβαίνουν σαφώς τα όρια που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη διπλή στήλη στην περιοχή Ρούντολφσπλατς και μετά στον αυτοκινητόδρομο του Τάουερν. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος τον Φεβρουάριο προσέφυγε για παραβίαση της συνθήκης κατά της Αυστρίας για μη τήρηση των προδιαγραφών της ε, ...ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Τι σημαίνουν τώρα αυτές οι ε, υψηλές τιμές. Οι τιμές αυτές είναι από το 1996, έχουν αλλάξει ποιοτικά πολλά πράγματα, όμως ό,τι αφορά τις συνολικές εκπομπές ρηπαντών, βρισκόμαστε περίπου στις ίδιες τιμές. Σας παραπέμπω στην πρώτη γραμμή και στις δύο τελευταίες γραμμές που βλέπετε εδώ στην διαφάνεια. Ο Δόκτωρ Γκέρτ Όμπερφελτ, ιατρός του Σάλτσπουργκ, θεωρεί ότι από αυτή την παραβίαση των ε, τιμών των ατμοσφαιρικών ρήπων, είναι βεβαίως μία μελέτη αυτή, ωστόσο βοηθεί να προσεγγίσουμε το θέμα. Στη βάση των μελετών αυτών, κατά πάσα πιθανότητα, είχαμε αναέτος μέχρι 140 πρώιμους θανάτους που θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί λόγω της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Υπενθυμίζω πόσο σημαντικό είναι το αυτοκίνητο, το ιδιωτικό αυτοκίνητο στο Σάλτσπουργκ ε, για την κάλυψη έστω και σύντομων διαδρομών. Τα ιατρικά προβλήματα που αναφέρονται εδώ έχουν κοστίσει πιθανώς και μέχρι 170 εκατομμύρια έμεσο ή άμεσο κόστος, δηλαδή σημαντικό ποσό. Επισημαίνω επίσης ότι εάν κάνουμε την ανάλυση σε παρόντα χρόνο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η μελέτη με τα σωματίδια, θα πρέπει να επαναληφθεί η μελέτη διότι είναι πιο ε, διευκρινής περισσότερα τα πράγματα από τη μελέτη με τις τιμές 1-2. Δεν είναι διαθέσιμη η μελέτη αυτή, γι' αυτό έχω προσφύγει στις παλές αυτές τιμές και περιλαμβάνω και την παραπομπή σχετικά με το κόστος στον ιατρικό τομέα που θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί. Το ίδιο όπως στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε κάθε δεύτερη κοινότητα, θα έλεγα, βλέπετε εδώ χάρτη του Ομοσπονδιακού Κρατηδίου και με κόκκινο βλέπετε όλους τους δρόμους όπου ο θόρυβος από την κυκλοφορία είναι πολύ υψηλός και υπάρχουν μετρήσεις σε δεσιμπέλ στη βάση των οποίων οφείλει να πει κανείς ότι έχουν επιπτώσεις στην υγεία. Εν συνόψη, αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικός αριθμός των κατοίκων του Σάλτσπουργκ και βεβαίως και για αυτού που θα εξυπηρετήσει στο βόρειο μέρος της Βαβαρίας κλπ. θα μπορέσουν, εφόσον δημιουργηθεί ο σιδηρόδρομος, να μειωθούν σημαντικά και η ατμοσφαιρική ρήπη και ο θόρυβο. Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η δημιουργία ενός καλού μέσου, μεταφορικού μέσου, που για μας και την δική μας περίπτωση είναι ένας αστικός και προαστιακός σιδηρόδρομος που τα σχέδια υπάρχουν ήδη από τη δεκαετία του 90 του περασμένου αιώνα. Έχω σχετική μελέτη και σας παραπέμπω και στα έγγραφα που σας έχω διαβιβάσει, σχετικά δηλαδή με την, έργα, με το, με την εργασία του ε, μηχανικού κυρίου Μπράντλε. Θα μπορούν να μεταφέρονται 60.000 επιβάτες ανά ημέρα και θα φτάσει μέχρι τις 180.000 σε ιστερότερη φάση. Εφόσον υλοποιηθεί το δίκτυο αυτό, εδώ βλέπετε στην διαφάνεια αυτή, για να μπορέσετε να έχετε μια εικόνα πώς θα κινηθεί η γραμμή αυτή, η σχεδιαζόμενη αυτή η γραμμή του δικτύου. Εάν υλοποιηθεί λοιπόν το δίκτυο αυτό, όχι μόνο θα υπάρξει αύξηση της κινητικότητας, και επομένως πολλοί θα εγκαταλείψουν εθελοντικώς τα αυτοκίνητα για να ε, πάνε στο, να πάρουν το τρένο, αλλά θα δημιουργηθούν και θέσεις απασχολήσεως. Με την μετακίνηση από το ιδιωτικό αυτοκίνητο στα δημόσια μέσα μεταφοράς και χωρίς κανένα εξαναγκαστικό μέτρο θα οδηγηθούμε σε μείωση των ε, ατμοσφαιρικών ρήπων, αλλά και σε μείωση του θορύβου. Επ' αυτού θέλω να σημειώσω ακόμη ότι στο Σάλτσπουργκ έχουμε ορεινές περιφέρειες και είμαστε στους πρόποδες των Άλπαιων, δηλαδή εξαρτώμεθα περισσότερο από τις αλλαγές του κλίματος που προέρχονται από την αναθέρμανση του παγκόσμιου κλίματος και είχαμε και πρόσφατα σημαντικές περιορισμένες μεν ε, γεωγραφικά ε, συνέπειες, είναι όμως και αυτές ένας λόγος που συνηγορεί υπέρ της ε, δημιουργίας του σιδηροδρόμου, για να επιτευχθεί δηλαδή καλύτερη προστασία του κλίματος. Έχω και στατιστική της ε, Αυστριακής Ένωσης Ασφαλιστών που δείχνει ότι θα εξοικονομηθούν εκατομμύρια ανά έτος από ε, την ε, αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας κλπ. Έτσι λοιπόν ο σιδηρόδρομος είναι σημαντικός για μας πρωτίστως για την βελτίωση του κλίματος με ταυτόχρονη διατήρηση και δυνατόν βελτίωση της κινητικότητας και βεβαίως με σημαντική εξοικονόμηση κόστους. Θα ολοκληρώσω με αυτά. Είχα και μερικά στοιχεία ακόμη, δεν θέλω όμως να σας επιβαρύνω περισσότερο. Δείχνω μόνο μια τελευταία εικόνα που ίσως σας δίνει μια εντύπωση ε, της ε, περιοχής για την οποία σας ομιλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Έχουμε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Προστασία του Περιβάλλοντος. Παρακαλώ. Ναι, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον αναφέροντα για τις ε, εξηγήσεις που μας έδωσε, που βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσες. Όσον αφορά την ε, οδηγία για την ηχορύπανση. Εδώ πρέπει να πούμε ότι όπως έχουμε ήδη εξηγήσει στη γραπτή μας απάντηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί βάσει αυτής της οδηγίας να ζητήσει από τις χώρες να υιοθετήσουν κάποια μέτρα, σαν και αυτά ε, που μας είπε ο αναφέρον. Δεν βλέπουμε λοιπόν να υπάρχει νομική βάση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάληψη μέτρων. Έρχομαι τώρα στην οδηγία για την ποιότητα του αέρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να ανησυχεί για τις υπερβάσεις όσον αφορά τα οξύδια του αζότου στην Αυστρία και συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες, ιδιαίτερα στο Σάλσπουργκ όπου είχαμε 15 ε, μικρογράμμα ένα κυβικό μέτρο. Οι μελέτες όμως προσπάθησαν να βρουν την πηγή και είναι οι μεταφορές από ό,τι φαίνεται. Είναι οι μεταφορές που συνεισφέρουν περισσότερο στην κατάσταση αυτή. Χρειάζονται λοιπόν τοπικά, περιφοριακά και σε εθνικό επίπεδο μέτρα από πλευρά της χώρας για να μπορέσει η Αυστρία να συμμορφωθεί με την οδηγία για την ποιότητα του αέρος. Όμως, η οδηγία αυτή απαιτεί αποτελέσματα, δηλαδή δεν πρέπει να υπερβαίνουμε κάποιες τιμές. Δεν απαιτεί όμως συγκεκριμένα μέσα ή την εφαρμογή συγκεκριμένων μέσων. Οπότε η επιλογή των μέσων απομένει θέμα των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να αποφανθεί για την επιλογή του ενός ή του άλλου μέτρου προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός. Όμως, από τα στοιχεία της Επιτροπής, οι ετήσιες τιμές, πράγματι το 2010 υπήρχε σημαντική υπέρβαση των τιμών και το 2014, που είναι και τελευταία χρονιά για την οποία έχουμε δεδομένα, μεταξύ άλλων και στο Σάλσπουργο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν κατέληξε ότι δεν τηρεί μία από τις υποχρεώσεις της βάση της οδηγίας αυτής η Αυστρία. Επιπλέον η οδηγία επιβάλλει στις χώρες ε, μέλη την περίοδο υπέρβασης των τιμών να την κρατήσουν όσο γίνεται πιο σύντομη. υπάρχει λοιπόν θέμα με την ε, ποιότητα του αέρα. Εξού και ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2016 προσφυγή ή επιπαραλήψη από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη Αυστρία. Καλύπτεται και το Σάλτσμπουργκ στην αγωγή αυτή. Η Αυστρία είπε ότι στα τέλη του 2000, Ιουνίου του 2016 περιμένει να υπάρξει βελτίωση και θα μας απαντήσει. Στο μεταξύ λαμβάνουμε υπόψη μας αυτά που είπε ο αναφέρον και θα τα έχουμε υπόψη μας και στην ανάλυση που θα κάνουμε της απάντησης της Αυστρίας και μετά θα δούμε τι άλλα βήματα θα αναλάβουμε. Επαναλαμβάνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να πετύσει από την Αυστρία να υλοποιήσει συγκεκριμένα μέτρα, να λάβει δηλαδή συγκεκριμένα μέτρα. Όμως η Αυστρία πρέπει να διαλέξει τα μέτρα εκείνα τα οποία θα έχουν σαν αποτέλεσμα την επίτευξη του στόχου, μεταξύ άλλων και για το Σάλτσμπουργκ. Αυτό ακριβώς είναι που προσπαθούμε να πετύχουμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο? Γι' αυτό παρακαλώ, ο κύριος Γιάρου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω και την ερώτηση για τους αναφερόμενους, γιατί εγώ ως αδαής, ας το πω έτσι, έχω βεβαίως επισκεφτεί συχνά το Σάλτσφουρ, που βρίσκονται, είναι μια θαυμάσια πόλη, ως αδαής όμως αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα υποδομών που υπάρχει εκεί. Και όποιος ενδιαφέρεται ας πάει να δει. Το Σάλτσπουργκ έχει βεβαίως τα προβλήματα αυτά που υπαγορεύει η γεωγραφική του θέση, ε, τα ρεύματα κυκλοφορίας. Δηλαδή στην ουσία η κατάσταση καλή για ένα τέτοιο έργο. Ε, το ζητάει. Το ερώτημά μου είναι τι πήγε άσχημα, δηλαδή ποιος, ε, ε, ποιος διαφωνεί, τέλος πάντων ποιος δεν θα καταφέρει να συνεννοηθεί μαζί σας. Μπορώ να φανταστώ ότι ο δήμαρχος του Σάλτσπουργκ ε, θα είναι σύμφωνος. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή ο δήμαρχος να είναι κατά. Πού μπορεί να κολλάει λοιπόν το ζήτημα, γιατί όπως είπα εγώ ως αδαής θεωρώ ότι είναι αυτονόητο ότι ένα τέτοιο έργο είναι σκόπιμο. Έρχεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει ότι όντω το Σάλτσπουργκ έχει πρόβλημα. και εν τέλει και προς το συμφέρον των ανθρώπων που κατοικούν εκεί. Το ελάχιστο λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε είναι να αναζητήσουμε εντατικά, να βρούμε πού βρίσκεται το πρόβλημα, ποιος διαφωνεί με ποιον και γιατί δεν προχωρεί. Αυτό με απασχολεί στην περίπτωση. Έχω γνωρίσει τους Αυστριακούς ως ανθρώπους θετικούς και, και που δουλεύουν για το καλό. Πού βρίσκεται το πρόβλημα. Πρόεδρος, άλλος κανείς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ο αναφερόμενος. Ευχαριστώ για τις τοποθετήσεις και για τις ερωτήσεις. Το πρόβλημα έγκυται στο ότι έχουμε πολιτικούς στον Δήμο και στην Περιφέρεια που παρόλο που το έργο έχει προχωρήσει στον σχεδιασμό δεν επιθυμούν να το προωθήσουν. Εξακολουθούν να ευνοούν την κυκλοφορία ιδιωτικών αυτοκινήτων. Ως συμπλήρωση η σύνταγμα του Ντίτσεν που ενδέχεται μάλιστα να ενταχθεί και στα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έργα που όμως εξυπηρετεί μια μικρή κοινότητα μόνο και όχι την ευρύτερη περιφέρεια. Εμείς έχουμε γράψει ξανά και ξανά στο ομοσπονδιακό μας κρατήδιο να εκμεταλλευτεί την μελέτη Radio που έχει ε, προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα και με συγχρηματοδότηση 500.000 ευρώ και όλες μας οι αναφορές στο κρατήδιο του Σάλτσμπουργκ δεν έφεραν αποτέλεσμα, γι' αυτό αποφασίσαμε να αποταθούμε στις Βρυξέλλες γιατί οι πολιτικοί μα μπορούσα να σα πω και ονόματα, λένε ότι είναι σωστό το έργο, αλλά δεν κάνουν τίποτα περισσότερο. Και ο Δήμαρχος Δόκτωρ μπορώ να σα φέρω και ανακοινοθέντα τύπου ε, των σιδηροδρόμων, τον θεωρεί αντίπαλο. Τοποθέτησε μάλιστα επικεφαλής του αρμόδιου οργάνου κάποιον ο οποίος είναι αντίθετος με το έργο. Και γι' αυτό και για τη βελτίωση του περιβάλλοντος αλλά και για τη βελτίωση της κινητικότητας αναζητούμε και εμείς συμμάχους όπου αυτό είναι δυνατό. Ευχαριστούμε μεν για την μελέτη, αλλά έχει χρηματοδοτήσει και άλλα έργα έχει χρηματοδοτήσει και άλλες μελέτες έργων η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο μέλλον δεν χρηματοδοτηθεί το έργο για το Σάλτσπουργκ, θα το κατανοήσουμε βεβαίω αν δεν υπάρχουν χρήματα, αλλά δεν μας ε, ενδιαφέρει να χρηματοδοτούνται μελέτες οι οποίες καταλήγουν στα σιτάρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκόλτ. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε το εξής για την ώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα. Διότι Δεν ακούτε. Έχει... Μικρόφωνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι υπάρχει παραβίαση και έχει ασκήσει σχετική προσφυγή. Ακούσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να διατηρήσει προτίθεται να απαντήσει μέχρι οι αρχές Ιουλίου να κρατήσουμε λοιπόν ανοιχτή την ε, αναφορά. Μπορούμε να υποβάλουμε ερώτηση και στον Δήμο Σάλτσμπουργκ και στην περιφέρεια να ρωτήσουμε πού ακριβώς έγκυται το πρόβλημα. Αναφέρομαι στην πρόταση του κύριου Γιάρ. Αν συμφωνείτε, μπορούμε λοιπόν να κάνουμε έτσι και να ολοκληρώσουμε εδώ το θέμα αυτό. Τώρα προχωρώ στο 12 της ημερησίας διατάξεως. Πρόκειται για Ιταλική αναφορά για την ποιότητα του αέρα στην Βενετία. Αναφορά 2288-14 Τζουζέπε Τάταρα. So, good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for having me here. Ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Εδώ εκπροσωπώ 7 μη κερδοσκοπικέ ε, οργανώσεις και τους πολίτες που έχουν συνυπογράψει την αναφορά αυτή που σας υποβάλαμε. Η αναφορά αυτή ε, βασίζεται σε διάφορα στοιχεία μεταξύ άλλων την παραβίαση της ε, οδηγίας του 2008-15 που έχει να κάνει με την κυκλοφορία στα ύδατα της Βενετίας. Εδώ έχετε τις διαφάνειες αυτές που σας δείχνουν πώς κυκλοφορούν τα πλοία εκεί. Είναι η μπλε γραμμή και υπάρχει και η κίτρινη γραμμή που είναι η εναλλακτική. Και η στατσιόνε μαρίτιμα της ε, Βενετίας που είναι πάρα πολύ κοντά στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Βενετίας. Δεν είναι απλώς ε, στη θάλασσα, είναι στη Λαγκούνα, δίπλα στο ιστορικό κέντρο της Βενετίας. Η αναφορά λέει ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση με τα άρθρα 6 και 7 όσον αφορά την τοποθεσία του κέντρου αυτού του θαλασσίου. Λέει ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση με τις οριακές τιμές του PM10 και ούτε και όσον αφορά τις οριακές τιμές του διοξιδίου του αζότου. Για το πρώτο, όσον αφορά το σημείο συγκέντρωσης των πλοίων. Υπάρχει ένα μόνο στο ιστορικό, στην ιστορική πόλη αυτή της ε, Βενετίας. με PM2,5, ενώ η οδηγία ζητάει να βασιζόμαστε στις πηγές κυκλοφορίας. Ονομάζεται Background Station. Η πραγματική έκθεση του τοπικού πληθυσμού και των 300 εκατομμυρίων τουριστών ε, της Βενετής καταλαβαίνετε ότι πλήττει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Αριστερά βλέπετε το κέντρο μέτρησης και την ε, μέτρηση σε άλλο σημείο. 2 Μαΐου είναι τέσσερις φορές παραπάνω από την πρώτη μέτρηση στο κανάλι Τζουντέκα. Είναι διαφορετικές οι μετρήσεις αυτές. Αριστερά και δείξα. Και εδώ πέρα πάλι βλέπετε την ίδια μέρα στο Σεν Τέλενα και βλέπετε ότι στη μία περίπτωση φορές παραπάνω από ότι στην άλλη. Ανάλογα με το αν είσαστε ανάντι και κατάντι κάθε φορά. Τώρα, όσον ε, αφορά το PM10 και το PM2,5. Υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στην κυκλοφορία των πλοίων και την ρήπανση, εννοείται, στις μετρήσεις. Εδώ έχετε μετρήσεις από τις λιμενικές αρχές, που είναι και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Και είναι σαφή ο συσχετισμός. Εδώ Μπορεί βέβαια να πει κανείς, «Ε, είναι περιορισμένη η ρήπανση. Μπορεί μισή ώρα να ανεβαίνει. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί τα κρουαζιερόπλια παραμένουν πολύ κοντά στις κατοικίες στην Βενετία, στο Σανταμάρο, με 1,8 τόνους καύσιμα την ώρα και μένουν 19 ώρες. Οπότε η κατανάλωση είναι 34 τόνοι ανασκάφος. Και στην ε, περίοδο μεγάλου τουρισμού έχουμε 5 με 7 τέτοια πλοία. Οπότε η κατανάλωση τόνων καυσίμων είναι 200 τόνοι περίπου την ημέρα. Το Σαββατοκύριακο το καλοκαίρι. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι τα χρησιμοποιούν συνέχεια καύσιμα τα σκάφη, το βλέπετε εδώ και όταν βρίσκονται δηλαδή εκεί στη Βενετία. Και εδώ πέρα βλέπετε τι ισχύει όσον αφορά το PM2,5 στην Βενετία, στο Άπιτσε. Είναι η τοπική υπηρεσία μέτρησης στο Άπιτσε και εξηγεί ότι το ίμιση της ρήπανσης οφείλεται στο λιμάνι, στα επιβατικά και εμπορικά σκάφη που περνούν από τα νερά εκεί. Το μισό της ρήπανσης ε, δηλαδή στην κοινότητα της Βενετίας οφείλεται ακριβώς αυτή την κυκλοφορία, τη θαλάσσια. Η εσωτερική, στα εσωτερικά ύδατα η μεταφορά επίση είναι ε, πολύ σημαντική και επιδεινώνει την ε, ρήπανση στο Ριάλτο, στη Γέφυρα για παράδειγμα όπως σε ένα τούνελ που βρίσκεται σε ένα μεγάλο αυτοκινητόδρομο. Μόνο που στους αυτοκινητοδρόμους και στα τούνελ τους δεν ζουν άνθρωποι, ενώ εδώ στην Βενετία ζει κόσμος και περνάνε εκατομμύρια τουρίστες. Μια εικόνα είναι αυτή που φαντάζομαι θα την ξέρετε, θα είστε εξοικειωμένοι με αυτή τη φωτογραφία. Τα βαπορέτο είναι επίσης υπεύθυνα για την ρήπανση της ατμόσφαιρας. Τώρα, ερχόμαστε στη μη συμμόρφωση με τις οριακές τιμές διοξιδίου του αζότου όσον αφορά την προστασία της ε, ανθρώπινης υγείας. Τα ξέρουμε αυτά, αλλά θέλω να πιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι η ρήπανση αυτή καταστρέφει και τα μνημεία. Είναι γνωστό το πώς, ε, τι πέτρα χρησιμοποιούμε που είναι ο στην Βενετία που χρησιμοποιείται για τη διακόσμηση μνημείων αλλά και για τα ίδια, τα δομικά τους τα υλικά, κολόνες κλπ. Και τα οξύδια αυτά, όπως επίσης δηλαδή και του αζότολ και του θείου, καταστρέφουν τα υλικά αυτά. Τα βλέπετε αυτά σε αυτές τις δύο φωτογραφίες και βλέπετε πόσο τα θικά οξύδια καταστρέφουν Τελικά αυτά και αυτά τα μνημεία. Το ανάγλυφο δηλαδή των ε, μνημείων αυτών. Τώρα, δεν έχει ληφθεί υπόψη κάποιο μέτρο προστασίας στο τοπικό σχέδιο και αυτό που ζητάμε εμείς να υπάρξει κοινοποίηση στην Ιταλική κυβέρνηση όσον αφορά τις περιπτώσεις που έχουν διαπιστωθεί τέτοια προβλήματα οι μετρήσεις που έχουν γίνει και για το PM5, αλλά και για το ότι χρειάζεται ένα υποχρεωτικό σχέδιο με χρήση φίλτρων, για παράδειγμα, ή άλλων ε, μηχανισμών, όπως συμβαίνει στις κανονικές πόλεις, εντό εγωγικών το κανονικές, για να αποφεύγονται οι επιπτώσεις από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Το ίδιο να γίνει και εδώ για τα πλοία, τα βαπορέτο, τα εμπορικά κλπ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Μάρτα Μουνιό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την DG Περιβάλλον. Θέλω να σα ευχαριστήσω για την πολύ χρήσιμη αυτή ε, εισήγηση. Δεν θα επαναλάβω την απάντηση που έχει ήδη δώσει τον Μάρτιο του 2016 η Κομισιόν, αλλά θα ενημερώσω για το εξελίξεις ε, σε σχέση με την έρευνα που έχει κάνει η Κομισιόν για το θέμα, ιδιαίτερα όσον αφορά τον αριθμό των σταθμών δειγματοληψίας ε, στην περιοχή της Βενετίας ε, καθώς και τη συμμόρφωση με την τοποθεσία των σταθμών δειγματοληψίας. Ε, ξεκινήσαμε μια, μια μελέτη για τον αριθμό των σταθμών δειγματοληψίας στην ζώνη της Βενετίας και φαίνεται να είναι συμβατός ο αριθμός των 108 σημείων είναι ε, αυτό συμβατό με τον αριθμό, με, το... με την κυκλοφορία. Φαίνεται λοιπόν να υπάρχει συμμόρφωση με τον ελάχιστο αριθμό δειγματοληπτικών σταθμών όπως απαιτείται από την ε, ε, οδηγία στο παράρτημα της οδηγίας. Η... Τώρα, όσον αφορά το πού βρίσκονται οι δειγματοληπτικοί σταθμοί, μετά από τις εξηγήσεις που λάβαμε, βλέπουμε ότι στην πράξη δεν συμμορφούνται η κατάσταση με την ε, οδηγία για την ποιότητα του αέρα. Στο τρίτο παράρτημα απαιτείται τα σημεία δειγματοληψίας να βρίσκονται εκεί όπου υπάρχει η μεγαλύτερη σώρευση και η μεγαλύτερη, η πιο μάλλον πυκνή ε, πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Επίσης, στο δεύτερο στο παράρτημα Β απαιτείται η εκτίμηση βιομηχανικών, ε, βιομηχανικής ρήπανσης ε, τουλάχιστον με ένα δειγματοληπτικό σταθμό ο οποίος θα πρέπει να βρίσκεται κατά του ανέμου. Από ό,τι φαίνεται αυτό δεν ισχύει οπότε θα μελετήσουμε περαιτέρω την κατάσταση για να δούμε αν πραγματικά υπάρχει παράβαση. των διατάξεων στην ιστορική πόλη της Βενετίας. Όταν οριστικοποιήσουμε την έρευνά μας θα αποφασίσουμε για τα περαιτέρω βήματα. Αυτά σε σχέση με την τοποθεσία για τον αριθμό των δημογματοληπτικών σταθμών. Τώρα, όσον αφορά τη διαδικασία κατά παράβαση, δεν μπορούμε να προσθέσουμε τώρα κάτι παραπάνω, γιατί ήδη αυτό το έχουμε εξηγήσει και στην απάντησή μας. Δεν ξέρω, μπορούμε κάτι να προσθέσουμε παραπάνω. Όχι. Αυτά ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Με ειδοποίησαν ότι υπάρχει εκπρόσωπος της Ιταλικής κυβερνήσεως. Έχετε το λόγο. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους. Όντως έχω κάποια στοιχεία που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας σε σχέση με την ποιότητα του αέρα στην Βενετία. Σύντομα να σας πω ότι η περιφέρεια του Βένετο έχει προβλέψει στο να, μοιράσει σε ζώνες την περιφέρεια σύμφωνα με το άρθρο 4 της ε, ε, οδηγία 2008-50 από τον Οκτώβριο του 2012. Η πόλη της Βενετίας στο πλαίσιο του διαχωρισμού εντάχθηκε στη ζώνη 508, δηλαδή αστική περιοχή της Βενετίας. Τα κριτήρια που ορίζονται από το 5ο και το 1ο παράρτημα της οδηγίας έχουν ε, ε, έτσι οριστεί συγκεκριμένα σταθερά σημεία δειγματοληψίας που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση ε, της περιοχής. Οι δειγματολογιστικοί σταθμοί λοιπόν ορίστηκαν από τις Ιταλικές Αρχές σύμφωνα με την τοποθεσία τους σε μικροκλίμακα και μακροκλίμακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 3 της Οδηγίας 2850. Όσον αφορά για τους σταθμούς για τον μέτρηση του όζοντος, που είναι η Φυσουόλα και η Σάκα Φίζολα, ορίστηκαν από το 8ο παράρτημα της Οδηγίας 2008-50, όπου προβλέπεται ρητά για τους ε, δηματοληπτικούς σταθμούς ε, αστικού τύπου τοποθεσία μακριά από την εισρωή τοπικών εκπομπών, όπως η κυκλοφορία ή... σταθμοί καυσίμων, έτσι ώστε να υπάρχει συγκεκριμένη ε, και εξασφαλισμένη κυκλοφορία αέρα. Να μην είναι κοντά δηλαδή σε δέντρα, να μην είναι κοντά σε πλατείες όπου δεν υπάρχει κίνηση, να μην είναι κοντά σε σχολικές ε, εγκαταστάσεις, σε εγκαταστάσεις αναψυχής ή παιδικές χαρές. Σύμφωνα με το παρακάτω παράρτημα, ο σιδηροδρομικός σταθμός ε, Μαργέρα θεωρείται ειδικά σταθμός που στη συγκεκριμένη περίπτωση της Βενετίας υπάρχει τόσο για να εξυπηρετεί το λιμάνι όσο και για τις εμπορικές δραστηριότητες. Ε, θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η βιομηχανική ζώνη Μαργκέρα Ε, έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των λιμενικών και αυτά όλα σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της Οδηγίας 2008-50. Ο Δήμος της Βενετίας εξάλλου έχει υποστεί σε επιπλέον ε, ελέγχους ε, για την βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου και της ε, Βενετίας αλλά και της περιφέρειας του Βένετο όσον αφορά την ναυτική κίνηση, την, μάλλον την κίνηση πλοίων στην Βενετία. Να θυμίσω δε και μια εκστρατεία ελέγχου με μετακινήσιμου σταθμού δείγματοληψία δίπλα στον ε, λιμάνι της Σάντα Μάρτα και ακόμα μια εκστρατεία με συγκεκριμένου κινητού σταθμού δείγματοληψία σε άλλε δύο συγκεκριμένες περιοχές τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Πέρα από αυτά, και για να έρθω σε πιο πρόσφατε ημερομηνίε, δεδομένου ότι η τελευταία απάντηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρονολογείται από το Μάρτιο του τρέχοντο έτου, να σα πω ότι τον Απρίλιο φέτο, το 2016, η περιφέρεια του Βένετο ενέκρινε ένα νέο περιφερειακό σχέδιο προστασία και ατμοσφαιρική εξυγίαση, που περιλαμβάνει συγκεκριμένε δράσει που έχει προγραμματίσει η συγκεκριμένη περιφέρεια μέχρι το 2020, ώστε να μειωθούν οι εκπομπέ και να γίνουν σεβαστές, σεβαστές οι τιμές που ορίζονται από την οδηγία του 2008. Αυτό το πρόγραμμα αφορά τις εκπομπές του λιμανιού αλλά και νέες δράσεις για τα λιμάνια από τις δράσεις α8.6 μέχρι 12α. Ανάμεσα σε αυτές τις δράσεις θα πρέπει ίσως να σας θυμίσω τη δράση που προβλέπει την ηλεκτροδότηση των ε, σταθμών ε, ηλεκτροδότησης ώστε να περιοριστεί η στάση των πλοίων στο λιμάνι ε, και κυρίως ε, θα έλεγα η τελευταία δράση είναι η Α812α που προβλέπει ένα σχέδιο παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα με κινητά εργαστήρια σε συνεργασία μεταξύ του Δήμου της Βενετίας και του Εθνικού της Εθνικής Υπηρεσίας ε, Προστασίας του Αέρα της περιοχής, της περιφέρειας μάλλον του Βένετο. Επίσης υπάρχει πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα με συγκεκριμένα σημεία που θα πρέπει να εντοπιστούν ε, σε συνεργασία με, την, ε, αυτό τον οργανισμό, τον περιφερειακό που σας ανέφερα για τον έλεγχο του αέρα. Ε, μάλιστα, οι λιμενικές αρχές της Βενετίας προχωρούν για να ορίσουν την τοποθεσία όπου, μαζί με τις λιμενικές αρχές όπου θα εγκατασταθεί ο νέος δειγματοληπτικός σταθμός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ε, κύριε. Επιθυμεί κανείς εκ των συναδέλφων. Ορίστε εσείς. Η ε, κυρία Εύη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε βρισκόμαστε ενώπιον ενό προβλήματο που είναι πραγματικά πολύ σοβαρό. Το πρόβλημα τη ποιότητα του αέρα σε ολόκληρη την Ευρώπη και όλο ιδιαίτερα σε ορισμένε περιφέρειε της Ευρώπης όπως αυτές της κοιλάδα του ΠΟ όπου έχουμε την περιφέρεια του Βένετο αλλά και της Λομβαρδίας που θα δούμε αργότερα με, ένα, με μια άλλη αναφορά για αυτό το θέμα είναι ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς ε, εξελίσσεται εδώ και πολλά χρόνια και που οι πολιτικοί και οι πολιτικοί ηθήνοντες δεν έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημα. Εγώ έχω την εντύπωση ότι για παράδειγμα σε σχέση με τα, τους σταθμούς μέτρησης ή δειγματοληπτικούς σταθμούς που, γίνονται, που αναφέρονται σε αυτή την ε, αναφορά φαίνεται να υπάρχουν πολύ διαφορετικές θέσεις. Οι αναφερόμενοι ανα... Ε, λένε πως η τοποθέτησή τους είναι τελείως ακατάλληλη και ότι δηλαδή δεν μετρά σωστά τα στοιχεία, ενώ η Ιταλική αντιπροσωπεία που την ευχαριστώ που βρίσκεται εδώ, χαίρομαι που βλέπω πως η Ιταλική αντιπροσωπεία συμμετέχει και παρακολουθεί ποιες είναι οι αναφορές που αφορούν την Ιταλία. Δεν μπορώ βέβαια να πω το ίδιο για το προηγούμενο, την προηγούμενη αναφορά όπου ήταν εξίσου σοβαρό το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, Υπάρχουν διαφορετικέ απόψει. Η Κομισιόν μα λέει όμω πω τρέχει η έρευνα και άρα θα αξιολογήσει αν και κατά πόσο υπάρχει παραβίαση, παράβαση. Συγγνώμη. Κατά εμά πρόκειται για προφανή παράβαση και ότι πρέπει να γίνουν συγκεκριμένε δράσει. Όμω η Ιταλία βρίσκεται σε μια κατάσταση μη συμμόρφωση και για άλλε ε, ε, οδηγίες που θίγονται εδώ μέσω των αναφορών. Και εγώ πρόσφατα έκανα μία ερώτηση ε, μαζί με άλλους συναδέλφους όπου η Κομισιόν και ο Επίτροπος Βέλα αναφέρονται στις τρέχουσες ε, έρευνες και επίσης ε, ότι μπορεί να μηνυθεί η Ιταλία, κυρίως για την καθυστέρηση με την οποία διαβιβάζει τα στοιχεία, τα σχετικά με την ποιότητα του αέρα σε σχέση με τα όρια της απαιτήσει της ευρωπαϊκής. Υπάρχουν πολλά που πρέπει ακόμα να γίνουν. Ο πολιτικός κόσμος έχει τεράστιες ευθύνε και φυσικά στην περίπτωση της Βενετίας πρέπει να ενεργήσουμε όσο γίνεται πιο σύντομα γιατί η ναυσιπλοεία και έχει τεράστιο αντίκτυπο στην υγεία των κατοίκων της πόλης και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Ε, θέλω λοιπόν να μην ανοιχτεί αυτή η αναφορά, να παρακολουθήσουμε σοβαρά ποια είναι τα προγράμματα που προτείνει η Ιταλία και η περιφέρεια του Βένετο για να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πέτερ Γιάρα. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτη, Χαίρομαι και ευχαριστώ που ήταν παρόν και εκπρόσωπος της κυβερνήσεως της ενδιαφερόμενης χώρας μέλους. Αυτό ας αποτελέσει παράδειγμα και για άλλους. Γνωρίζω βεβαίως ότι συχνά προσκαλούνται, αλλά ότι σπανίως λαμβάνουν τον κόπο να προσέλθουν. Με τον τρόπο αυτό όμως γίνεται και καλύτερος διάλογος. Δεύτερο, θα συμφωνήσω με την προγραλή σας να μην ανοιχτεί η αναφορά από όσο κατάλαβα υπάρχουν δύο προβλήματα. Μπορεί κανείς βέβαια να διαφωνήσει για το πού θα πρέπει να εγκατασταθούν οι μονάδες μετρήσεως. Αυτό που φαίνεται ωστόσο αδιαμφισβήτητο είναι ότι οι μετρήσεις δείχνουν τιμές άνω των επιτρεπομένων. Αναμένω λοιπόν από τη χώρα μέλος, την Ιταλία δηλαδή, να λάβει μέτρα. Γνωρίζω ότι η κίνηση των σκαφών αυτών γίνεται με πεπαλαιωμένες μηχανές δίζελ. Χρειάζεται να ληφθεί μέρημνα λοιπόν, να αντικατασταθούν. Γνωρίζω ότι υπάρχει και συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τα αυτοκίνητα υπάρχουν και καταλήτες βεβαίως. Για τα πλοία, ωστόσο συνήθως δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόβλεψη. Τροφοδοτούνται και με ε, κακής ποιότητα καύσιμο, πολύ συχνά, ε, οι μηχανές δίζελ των ε, σκαφών. Ωστόσο δεν είναι μονάχα πρόβλημα της Βενετίας αυτό, να είστε σίγουροι. Απαντά και αλλού. Και όλα αυτά συμβάλλουν στην επιδείνωση της ατμοσφαιρικής της ποιότητας, δηλαδή του ατμοσφαιρικού αέρα. Να μην ανοιχτεί η αναφορά και βεβαίω ε, να αναζητηθούν οι αιτίε. Το πρόβλημα είναι βεβαίω γνωστό. Είναι, ο τουρισμός είναι καλός, αλλά πρέπει να λυθεί μέρημνα να μετακινούνται οι τουρίστες με κατάλληλο τρόπο. Ευχαριστώ. άλλο κανεί επιθυμεί να λάβει τον λόγο. Κύριε Τάτερα, εσείς λοιπόν μπορείτε να ολοκληρώσετε. Εκτός μικροφώνου μιλητής. Ναι, έχω κάποιες παρατηρήσεις να κάνω. Είναι αλήθεια ότι έχουν γίνει εκστρατείε με κινητούς σταθμούς ε, μέτρησης και όταν γίνανε αυτές οι εκστρατείε, ήταν πολύ περιορισμένες χρονικά, διαπιστώσαμε όντως πολύ διαφορετικές μετρήσεις από ότι η σταθερή σταθμή της ΣΑΚΑ Φίζολε. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο που στηρίζει την ε, αναφορά μας. Ε, εμείς δεν θέλουμε να έχουμε σταθερούς μόνο σταθμούς μέτρησης που να είναι κατάντι του αέρα και όχι ανάντι Έχουν γίνει μετρήσεις στους κήπους διαφόρων ξενοδοχείων και εκεί βλέπουμε ε, ε, την, τις μετρήσεις που είναι τουλάχιστον το διπλάσιο από ό,τι στην Σάκα Φίζολη, που δεν ζει κανείς στο συγκεκριμένο σταθμό μέτρησης, μόνο πουλάκια και εκεί. Ε, ε, δεν μετρώνται επίσης ούτε τα μεγάλα ε, τα ούτε τα μεγάλα εμπορικά πλοία. Δεν έχει μειωθεί καθόλου η ναυσιπλοεία, αντίθως έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και έτσι ε, ε, προτάθηκε και το να τοποθετηθεί ένα σταθμό μέτρη στη Φουζίνα. Ήταν μάλιστα αποτυχία αυτό γιατί εκεί υπήρχε πολύ μικρή κίνηση. Είναι ένα πολύ μικρό λιμάνι, το οποίο είναι λιματικό, άρα δεν χρησιμεύει σε κάτι να μετράμε ε, την ποιότητα του αέρα εκεί όπου μειώνεται η κυκλοφορία. Τώρα, Υπάρχουν λοιπόν κινητοί σταθμοί μέτρηση θα πρέπει να τοποθετηθούν πιο κοντά στην πόλη της Βενετίας που μάλιστα δεν μπορεί να εξετάζεται με, επί τη βάση των κατοίκων της μόνο, αλλά επί τη βάση τη μόνιμη τουριστική παρουσία, που ξέρετε ότι είναι τεράστια, ίσως και υπερβολική σε κάποιες χρονικές περιόδου. Ε, και δεν γνωρίζουμε κατά πόσο ο ηλεκτρισμός θα παρέχεται από το κεντρικό σταθμό της Μαργκέρα, ίσως καίγοντας, καίγοντας άνθρακα ή άλλες ή άλλα καύσιμα τα οποία ρηπαίνουν και πάλι πολύ την ατμόσφαιρα. Επαναλαμβάνω ότι οι επιθεωρήσεις και οι μετρήσεις θα πρέπει να δημοσιεύονται. Οι πλατφόρμες και οι σταθμοί μέτρησης να τοποθετούνται σωστά και οι άνθρωποι που ζουν στην πόλη αλλά και οι τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη μας να μπορούν να αναπνέουν καθαρό αέρα σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι ενισχύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτή είναι η κατάσταση, ναι, το πρόβλημα σαφώς και υπάρχει. Το αναγνωρίζει και η Επιτροπή και δουλεύει πάνω σε αυτό. Και η Ιταλία θέλει να συνεργαστεί. Κάτι το οποίο είναι θετικό, γιατί έτσι θα φτάσουμε πιο εύκολα στη λύση. Λοιπόν, πρέπει να δούμε το αποτέλεσμα όλων αυτών. Συνεπώς παραμένει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Συμφωνείτε? Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Και περνάμε τώρα στη, στο επόμενο σημείο. Είναι το σημείο 13 στην σε διάταξη. Πρόκειται για δύο αναφορές και οι δύο Ιταλικές. Άννα Γκερομέτα είναι η πρώτη αναφέρουσα. Και ο Ραφέλ Μπελέτσα, ο δεύτερος. Είναι η Άννα Γκερομέτα εδώ παρούσα, έτσι, για να μας παρουσιάσει την αναφορά της. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Θα σας διαβάσω αυτό που έχω ετοιμάσει. Αγαπητοί κύριοι, όταν στείλαμε επιστολή το 2013 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητώντα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει νέα δράση σε βάρος της Ιταλίας η οποία δεν τηρεί τα όρια για τη ρήπανση του αέρα βάσει της οδηγίας για την ρήπανση του αέρα θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι μετά την ε, απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 2012 που καταδίκασε την ε, Ιταλία επειδή παραβίαζε τα όρια του PM10, θα στέλναμε ένα σαφές μήνυμα προς τις κυβερνήσεις μας, ότι οι κανόνες δηλαδή για την ποιότητα του αέρα προστατεύει όντως τον πληθυσμό από την ρήπαση του αέρος και άρα πρόκειται για μια προτεραιότητα που δεν πρέπει να παραβιάζεται. Εδώ τώρα ανανεώνω το έτοιμά μου και επαναλαμβάνω ότι πρέπει να ληφθεί επιγόντως δράση προκειμένου να ισχύει ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποιότητα του αέρος. Από το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νέα μέτρα σε βάρος της Ιταλίας για την παραβίαση των ορίων του PM10. Μία δράση η οποία όμως δεν συμπεριλαμβάνει όλες τις περιοχές που παραβιάζουν τα όρια για την ποιότητα του αέρος. Γιατί αποκλεί τις περιοχές εκείνες οι οποίες πρόσφατα έχουν εκδώσει σχέδια για την προστασία ε, του αέρα, αλλά που δεν έχουν τηρήσει ακόμα τους στόχους έτσι όπως αυτοί προβλέπονται από την οδηγία για την ε, ποιότητα του αέρος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο το όλο εγχείρημα, γιατί έτσι δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη οι περιφερειακέ αρχέ και στέλνεται και ένα λάθο μήνυμα προ τι κυβερνήσει, λε και τελικά το θέμα τη ποιότητα του αέρα είναι κάτι το οποίο μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Ξεκινώντα λοιπόν με τη δράση αυτή για το PM10, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πίστεψε ότι έτσι θα συμπεριλαμβάνονταν μέτρα τα οποία θα άλλαζαν την κατάσταση. Δεν έγινε όμως αυτό και έτσι η παραβιάση, η δράση μάλλον κατά της Ιταλίας για την παραβίαση του PM10 πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις περιοχές που εξακολουθούν να παραβιάζουν την οδηγία αυτή. Δεδομένου ότι οι παραβιάσεις αυτές όσον αφορά τα όρια συνεχίζεται και πάρα πολύ καιρό, τη δράση αυτή, όπως εκείνη και για το διοξίδιο του αζότου, πρέπει να την ισχύσει ακόμα περισσότερο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να υποχρεώσει τις χώρες να προχωρήσουν στην υλοποίηση των σχεδίων που έχουν προβλέψει. Η Λομβαρδία, για παράδειγμα, είναι μία από τις περιοχές που έχει τις χειρότερες συνθήκες όσον αφορά την ποιότητα του αέρου, γιατί υπερβαίνει τις ε, οριακές τιμές και για το PM10 και για το PM2,5 και για το όζον ε, και για το βάριο πι, για το διοξίδιο του αζότου. Και η γεωγραφική θέση είναι τέτοια που πρέπει να γίνουν επιπλέον προσπάθειες για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί εκεί από ό,τι αλλού. Τα μέτρα όμως πρέπει να είναι τέτοια που να έχουν αποτέλεσμα, να έχουν και κατάλληλη χρηματοδότηση και να ελοποιούνται επιγόντως έτσι ώστε να προστατεύεται η υγεία των πολιτών. Όσον αφορά τώρα το περιφερειακό έδρος για το σχεδιασμό, ε, την προστασία όσον αφορά την ποιότητα του αέρου στην Λομβαρδία. Στόχος είναι να προστατευτεί η υγεία βέβαια των πολιτών. Το 2015 όμως 100 φορές είχε υπερβεί τα ημερήσια όρια για το PM10 η Λοβαρδία. 40 φορές παραπάνω από ότι το 2014. Συνεπώς πρέπει να υπάρχουν προτεραιότητες και αποφασιστικότητα που δεν υπάρχουν σήμερα. Το 2014 αφού εγκρίθηκε σχέδιο το οποίο προβλέπει να καταργηθούν τα διτροχαπηδή είναι αυτά τα οποία ρηπαίνουν περισσότερο, η Λοβαρδία αποφάσισε να επιδοτήσει 350.000 τέτοια οχήματα. Μαζί με κάτι μίνι οχήματα, τα περισσότερα από τα οποία έχουν οι κινητήρες που λειτουργούν με δίζελ. 10 εκατομμύρια λοιπόν ήταν η απώλεια αυτή για την περιοχή, ενώ θα μπορούσε έτσι να έχει χρηματοδοτήσει 800 ηλεκτρικά ε, οχήματα για τις αστικές ε, περιοχές και να μειωθεί έτσι η ρήπανση του αέρα στη Λοβαρδία. Έστω σε ένα βαθμό, αλλά καλύτερο από το τίποτα. Το... Η έκθεση όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου για την ποιότητα του αέρος του 2015 λέει ότι πολλά από τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν εξαιτία της έλλειψης χρηματοδότησης. Άρα οι προσπάθειες της περιοχής για την ε, προστασία της ποιότητας του αέρα είναι πραγματικά κάτω από το 1% σε σχέση με το συνολικό προπολογισμό. Το 2015 δεν εγκρίθηκαν μέτρα από την περιφερειακή κυβέρνηση, το οποίο δείχνει ότι τελικά δεν υπάρχουν νέα σχέδια για να αντιμετωπιστεί κάτι το οποίο ήταν γνωστό ότι θα προκύψει στην Λομβαρδία. Η πίεση προς την Ευρωπαϊκή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την τοπική κυβέρνηση βοήθησε κάπως να υπάρξει μια σχετική οδηγία που λέει ότι τα μέτρα πρέπει να υλοποιηθούν και να έχουν αποτελέσματα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Όμως το 2015 οι περισσότερες περιοχές που βρίσκονται στην κοιλάδα του ΠΟ είχαν τέτοιες περιπτώσεις υπέρβασης των οριακών τιμών. Και αυτό το λένε και όλοι οι εμπειρογνώμονες. Το 2013 οι περιφερειακές κυβερνήσεις της κοιλάδας του ΠΟ και τα κύρια Υπουργεία υπέγραψαν μια συμφωνία προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να πνέουν καθαρό αέρα. Όμως τρία χρόνια μετά η συμφωνία αυτή έπρεπε να ήταν αυτό το οποίο θα άλλαζε την κατάσταση όσον αφορά την ποιότητα του αέρα στην κοιλάδα του ΠΟ, χωρίς όμως κανένα απολύτω αποτέλεσμα. Δεν έχει αλλάξει ούτε η πολιτική, ούτε έχουν εγκριθεί μέτρα και το συμπέρασμα λέει ότι 65% και πάνω από 35.000 πρώιμους θανάτους ε, έχουμε το χρόνο στην κοιλάδα του ΠΟ, στις περιοχές αυτές που βρίσκονται στην κοιλάδα του ΠΟ. Εδώ βλέπετε σε εθνικό επίπεδο τι γίνεται στη διαφάνεια αυτά. Η μείωση έχει να κάνει των οριακών τιμών, δηλαδή απλώς και μόνο με την κρίση και όχι με πολιτικές που έχουν τεθεί σε εφαρμογή και ότι το 2020 θα έχουν ε, αυξηθεί και πάλι οι τιμές, πολύ πάνω από τις οριακές. Εδώ στις μικρές διαφάνειες βλέπετε πώς ήταν ο αέρας το 2010 και δίπλα το 2020 αν η νομοθεσία συνεχιστεί ως έχει τώρα. Η ποιότητα του αέρα δηλαδή, κυρίως στη Βενετία, θα χειροτερέψει. Τέλος, Εξαιτία τη κρίση ε, με την ρήπανση του έρωτου του 2015, το Υπουργείο Περιβάλλοντος αποφάσισε με τις περιφερειακές ε, κυβερνήσεις νέα, ε, μη δεσμευτικά όμω μέτρα για τις μελλοντικέ πολιτικές. Με ελάχιστη όμως χρηματοδότηση ω καθόλου και μερικές φορέ τα μέτρα αυτά είναι λιγότερο αυστηρά από τι πολιτικέ που ήδη ισχύουν σε μερικέ περιοχέ τη χώρα σήμερα. Για παράδειγμα, το Ιταλικό Κοινοβούλιο εγκρίνει ένα σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας εθνικό με 35 εκατομμύρια για 46 πόλεις. Αυτές οι πόλεις λοιπόν Ιταλικές με τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα πώς θα βελτιώσουν την κινητικότητα με λιγότερο από ένα εκατομμύριο η καθεμία. Αν τα χρήματα φτάναν ίσως αν είχαμε μια βρύση που έτρεχε χρήμα. Αλλά τώρα πώς είναι δυνατόν να υλοποιηθούν σε ολόκληρη την Ιταλία τέτοια σχέδια κινητικότητες. Η Ιταλία λοιπόν εντελώ τυχαία αποφασίζει για κάποια μέτρα. Αν είμαστε σοβαροί για να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα για όλους τους Ιταλούς, τότε θα έπρεπε να αλλάξουν πολλά. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί Ευρωβουλευτές, βασιζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξει το έτοιμά μας για ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας του αέρα που αναπνέουμε. Και τελειώνω με το εξή. Επιμένουμε στην αναφορά μας και θέλουμε η Ιταλική κυβέρνηση να κληθεί να υλοποιήσει με επαρκή χρηματοδότηση τα μέτρα για την προστασία του αέρα σε συμμόρφωση με το άρθρο 23 της Οδηγίας για την Ποιότητα του Αέρα. Οι τιμέ πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο χαμηλές και αυτό να επιτευχθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρος. Έχουμε διαθέσιμους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να σας κάνω μια ενημέρωση για την κατάσταση η τελευταία ανακοίνωση της Επιτροπής είναι το Νοεμβρίου 2014. Για το 5, στο σημείο 5 δηλαδή, αναφέρεστε σε τιμή η οποία αναφέρεται μόνο στο 2015. Μάλλον στο 2014, ενώ τα ε, δεδομένα του 2015 δεν υπάρχουν ακόμα. Δεν μπορούμε λοιπόν να επαληθεύσουμε τα έχει μπερδέψει λίγο με τις χρονολογίες. 2016 εννοώ, μόνο, μόνο τότε, 2016, τέλος το 2016 θα έχουμε τα δεδομένα για να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε τις υπερβάσεις των τιμών. Τώρα, όπως είπατε στην πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας, για την οποία σα ευχαριστώ πολύ, επιστολή, επίσημη επιστολή εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2014 και όπως είπαμε στην επιστολή αυτή αναφερθήκαμε σε θέματα ε, ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα, παραβιάσεων της οδηγίας. Δεν είχαν περιληφθεί ορισμένες περιφέρειες της κοιλάδας του ΠΟ και ο λόγος για τον οποίο δεν περιλήφθηκαν οι περιφέρειες αυτές ήταν διότι είχαν πολύ πρόσφατα εγκριθεί σχετικές τιμές και τα σχέδια και έπρεπε να εξετάσει τα σχέδια αυτά σε βάθο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν να αποφασίσει για τι περιφέρειες αυτέ. Μπορώ να σα πω λοιπόν το εξή. Έχει ήδη αξιολογήσει τα μέτρα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαπιστώσαμε δε ότι τα μέτρα που προτείνει η Ιταλική κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν είναι επαρκή τα μέτρα και θα ακολουθήσουν επόμενα βήματα. Πολύ σύντομα. Αυτό μπορώ να σας το ανακοινώσω ήδη από σήμερα σε ό,τι αφορά το οξύδιο του αζότου. Επίσης στάλθηκε επιστολή στις Ιταλικές Αρχές το Μάιο του 2015 για την υπέρβαση των τιμών του οξυδίου του αζότου για διάφορες περιφέρειες και σε, σύμφωνα με το άρθρο 13 και το άρθρο 23 ότι δηλαδή δεν είχαν γίνει επαρκείς μετρήσεις για να είναι το δυνατόν συντομότερες οι περίοδοι υπέρβασης των ορίων. Σε σχέση λοιπόν με τις εκθέσεις ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα θα προχωρήσουμε σε επόμενα μέτρα. Με την άδειά σας τώρα κύριε Πρόεδρε θα μου επιτρέψετε να περάσω το μικρόφωνο στον συνάδελφό μου της ε, μονάδας ε, προσφυγών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, που δίνετε την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει στην αναφορά. Γνωρίζουμε το μέγεθος του προβλήματος των 20 εκατομμυρίων ανθρώπων που εκτίθενται στην κοιλάδα του ΠΟ σε αυτές τις υπερβάσεις των τιμών των PM10. Μετά από την απόφαση να στραφούμε κατά Πολωνίας και Βουλγαρίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έχουμε δύο υποθέσεις ήδη για υπέρβαση των ε, οριακών τιμών των PM10, κάτι που είναι σαφές από τα πιο πρόσφατα δεδομένα, έστω και αν δεν έχει γίνει ακόμη η επισήμωση αξιολόγησή τους, είναι ότι ο αριθμός των υπερβάσεων στην Ιταλία το 2015 δείχνει σαφώς μια φθήνουσα τάση, η οποία έχει σταματήσει. Η φθήνουσα ε, τάση έχει σταματήσει για τα PM10. Φαίνεται αυτό ωστόσο να οφειλόταν, η φθήνουσα τάση δηλαδή, σε ευνοϊκές μετεωρολογικές συνθήκες και όχι σε μέτρα που έλαβαν οι θυγόμενες περιφέρειες. Γι' αυτό μπορείτε να στηρίζεστε σίγουρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αξιότιμοι ευρωβουλευτές αλλά και αξιότιμοι αναφερόμενοι, διότι θα πράξουμε αυτά που κάναμε και κατά Βουλγαρίας και Πολωνίας, διότι πρέπει να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση, όπου δηλαδή αναφύονται παρόμοιε υποθέσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με όμοιο τρόπο. Ευχαριστώ. τα Ταβανάρη, έχετε το λόγο. E Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή. Η μόνιμη αντιπροσωπεία είναι σε διαρκή διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλες τις υποθέσεις που αφορούν ε, ε, διαδικασίες ε, κατά παράβαση σε σχέση με το περιβάλλον και θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να θυμίσω ότι η μόνιμη αντιπροσωπεία είναι πάντοτε παρούσα ε, κάθε φορά που καλείται σε συζητήσεις ε, της Επιτροπής για τις διάφορες αναφορές. Να θυμίσω μόνο ότι το τελευταίο 1,5 μήνα συμμετείχα και στην Επιτροπή για τις υποθέσεις διαχείρισης αποβλήτων ε, στο, στο Λάτσιο και για την υπόθεση ε, Ήλβα. Ήμασταν επίσης εδώ στη διάρκεια της προηγούμενης συζήτηση για την αναφορά για την γραμμή υψηλής ταχύτητας το Ρήνο Λιών, αλλά δεν εκρήθη απαραίτητο να παρέμβουμε στη διάρκεια εκείνης της συζήτησης και την αυτοαπόφαση της Ιταλικής κυβέρνησης δεν ήταν τυχαίο. Όσον αφορά τώρα τις συγκεκριμένες αναφορές για την ποιότητα του αέρα εν γίνε στη λεκάνη της ε, Παδανίας και στη Λομβαρδία, αυτό, οι παρατηρήσεις που μπορώ να κάνω και που μπορώ μπορεί κάπως να χρησιμεύσουν για την Επιτροπή σας. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να ενημερώσω για τις τελευταίες δραστηριότητες και τις δράσεις που έχουμε αναλάβει σε εθνικό επίπεδο. Συγκεκριμένα θα ήθελα να σας αναφέρω το γεγονός ότι όλες οι εργασίες ομάδων που έχουν δημιουργηθεί στο εσωτερικό του πλαισίου για το πρόγραμμα για την εξυγίανση της ατμόσφαιρας στη λεκάνη του ε, ΠΟ έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015 και στις αρχές 2016. Πρόκειται για 10 ομάδες εργασίας που αντιμετώπισαν, εξέτασαν μάλλον διάφορα θέματα περιβαλλοντικά ε, θέματα μεταφορών, θέματα γεωργίας. Να θυμίσω κάποια από αυτές τις ομάδες εργασίας στο εσωτερικό του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Έγινε, ε, ας πούμε, ε, μια στρογγυλή τράπεζα όσον αφορά τις πηγές δημιουργίας θέρμασης, θερμότητας μάλλον, μια άλλη, οι συζητήσεις ολοκληρώθηκαν στα τέλη του 2015 και ήδη έχουμε επεξεργαστεί σχετικό διάταγμα. Έχει σταλεί στα αρμόδια Υπουργείο και περιμένουμε να συντονιστούν τα αρμόδια Υπουργεία για να υιοθετήσουν αυτό το διάταγμα. Το ίδιο μπορούμε να πούμε για τη δεύτερη ομάδα εργασίας που ασχολήθηκε με την ενημέρωση των ανώτατων ορίων εκπομπών των εργοστασίων βιομάζας. Και εδώ συζητήσαμε συζητήσαμε για το... και καταλήξαμε σε διάταγμα και αυτό το διάταγμα έχει εκπονηθεί και είναι υποανάλυση από τους αρμόδιους υπουργούς ώστε να ε, οριστούν νέα κατάλληλα όρια για τα εργοστάσια που τροφοδοτούνται ε, από βιομάζα. Να θυμίσω και άλλες ε, τράπεζες εργασίας, ομάδες εργασίας που έκαναν βασική δουλειά γιατί ανάλυσαν πτυχές κρίσιμες ομάδα εργασίας που δημιουργήθηκε στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών είχε ως στόχο να ενημερώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τα ανανέωση των αστικών σχεδίων κινητικότητας. Αυτή η ομάδα εργασίας συνεργάστηκε και με την ομάδα εκπροσώπων των Ιταλικών Δήμων ακριβώς για να λάβει, ληφθούν έτσι υπόψη όλα τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις μεταφορές στις Ιταλικές πόλεις. Μια άλλη ε, ομάδα εργασίας ασχολήθηκε μέσα στο Υπουργείο Γεωργίας, Διατροφής και Δασών ασχολήθηκε με μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών από την γεωργία και την κτηνοτροφία. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις εργασίες που σας είπα ότι έγιναν με τα διάφορες, τις διάφορες ομάδες εργασίες για την λεκάνη της Παδανίας. Εξίσου συντάχθηκε ένα πρωτόκολλο συνεννόησης για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα ώστε να μην παροτρινθεί η χρήση των ιδιωτικών μέσων μεταφορών, μέτρα ώστε να προαχθεί η ενεργειακή επάρκεια, η χρήση ανανεώσιμων πηγών και ούτω καθεξής. Αυτό το πρωτόκολλο που ολοκληρώθηκε το 2015 προβλέπεται και έχει υπογραφεί μάλιστα αυτή τη στιγμή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος που είναι υπεύθυνο φυσικά για το θέμα σε εθνικό επίπεδο, όσο και από το κέντρο, το, και από τον πρόεδρο μάλλον της Ένωσης Ένωσης ε, ε, Περιφερειών αλλά και από το πρόεδρο της Ένωσης Δημάρχων της Ιταλίας. Ε, στις 30 Δεκεμβρίου 2015 υπήρξε συνάντηση ανάμεσα στους δημάρχους των μεγάλων αστικών κέντρων της Ιταλίας στην Ρώμη όπου συζητήθηκαν όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα του αέρα για όλη την επικράτεια την Ιταλική και εκεί έγινε μια συζήτηση κατά του νέφους ε, ανάμεσα στους υπουργούς και πιστεύουμε ότι μέσα στους επόμενες δύο εβδομάδες θα γίνει άλλη μια συζήτηση ανάμεσα στους προέδρους ε, των, και τους, ε, των, των περιφερειών και τους δημάρχους των μεγάλων αστικών κέντρων της Ιταλίας για τον ίδιο σκοπό. Εκεί όπου υπάρχουν ανοιχτές υποθέσεις και διαδικασίες παράβασης, γίνεται διάλογος και μπορώ να το πω αυτό γιατί είμαι ο άνθρωπος που ασχολείται με όλες τις διαδικασίες ε, κατά παράβαση ε, για θέματα που αφορούν το περιβάλλον στη μόνιμη ε, Ιταλική Αντιπροσωπεία. Υπάρχει καθημερινή επαφή με την Κομισιόν για όλες τις υποθέσεις που έχουν να κάνουν με παράβαση του κοινοτικού, της κοινοτικής νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ταβερνάρη. Η κυρία Εύη. Έχω μόνο μια σύντομη παρατήρηση. Σας παρακαλώ όλες και όλους να μιλάτε πιο αργά για να μπορούν να σας παρακολουθούν οι μεταφραστές. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κνέου. έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση, να εξετάσουμε μάλλον μια κατάσταση πολύ περίπλοκη. Λόγω των μορφολογικών και κλιματικών χαρακτηριστικών της λεκάνης της Παδανίας, ε, είναι η ε, ε, επειδή ακριβώς επικρατούν αυτές οι γεωγραφικές και μορφολογικές, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε αυτή την κατάσταση, τα προγράμματα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή δεν αρκούν. Μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο πλήττει εκατομμύρια κόσμο. Ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντο στην έκθεσή του τη περασμένη χρονιά μιλά για 450.000 πρώιμου θανάτου λόγω τη ε, ατμοσφαιρική ρήπανση. Στην Ιταλία αντιστοιχεί αυτό σε 84.000 ανθρώπου ετησίω. Προφανώ ε, είναι σοβαρότατο το πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλά με πνευματική ετοιμότητα. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει ούτε από πλευρά των τοπικών και εθνικών κυβερνήσεων, αλλά ούτε και από πλευρά τη Ευρώπη. Και εγώ εδώ στρέφομαι επίση και είμαι ευτυχή που είναι εδώ και η μόνιμη αντιπροσωπεία τη Ιταλία για να κάνω μια έκκληση. Έκκληση όσον αφορά τη διαπραγμάτευση για την οδηγία ΝΕΚ που σχετίζεται με τα εθνικά όρια εκπομπών. Γιατί, για παράδειγμα, η Ιταλία θα πρέπει να στηρίξει μια θέση για την προστασία της υγείας και όχι μείωση των ορίων που προβλέπονται μέχρι σήμερα και που είναι υπό διαπραγμάτευση. Θα πρέπει να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι θέλουμε πραγματικά να ενεργήσουμε για να προστατεύσουμε την υγεία των ανθρώπων και όχι απλά να μείνουμε στα νούμερα που μένουν απλά νούμερα στο χαρτί ή σε μηχανισμούς εικονικούς για να μπορεί να βασίζεται σε αυτά τα νούμερα η Κομισιόν όπως ας πούμε σήμερα για το ETS την εμπορία δηλαδή εκπομπών ένας μηχανισμός που βρίσκεται μόνο στα χαρτιά μόνο εικονικός είναι αυτός ο μηχανισμός και μόνο εικονικά προσπαθεί να περιορίσει τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα αλλά στην πράξη δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο γίνεται λόγος για μια διαφορά όσον αφορά την μείωση των εκπομπών όπως προτείνονται από την οδηγία ΝΕΚ για 15.000 ανθρώπους. 15.000 άνθρωποι μπορεί να χάσουν πρώιμα τη ζωή τους με βάση μάλλον αν γίνει η αλλαγή αυτή των ε, αριθμών, των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας και Επίσης και χαίρομαι που αναφέρθηκε το γεγονός ότι η γεωργία συμβάλλει επιδεινώνει την ατμοσφαιρική ρήπανση και εδώ καλό και πάλι την Ιταλία αλλά και όλα τα κράτη-μέλη που διαπραγματεύονται να μην αφαιρέσουν το μεθάνιο από τους ρήπους που πρέπει να παρακολουθούνται και να μειωθούν γιατί προφανώς αυτό θα σήμαινε μεγάλη ζημιά για την υγεία, τη δημόσια υγεία. Εγώ ως πολίτης που ζει στο Μιλάνο, κατοικώ στο Μιλάνο, έχω μεγαλώσει στο Μιλάνο και γνωρίζω πάρα πολύ καλά την περιοχή και πώς στη διάρκεια των ετών γίνανε επενδύσεις που ακολουθούν τελείως διαφορετική κατεύθυνση σε σχέση με τις ε, αντί για επενδύσεις για την προώθηση των ε, δημοσίων μεταφορών ενώ αντιθέτως, θα έπρεπε, ενώ αντιθέτως είδαμε να πολλαπλασιάζονται οι δρόμοι. Δεν λύνουν το, δε, το πρόβλημα της κίνησης, αντίθετα το επιθυνώνουν. Σε πολλά μέτωπα λοιπόν χρειάζεται περισσότερο θάρρος για ζητήματα που αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας, γιατί διαφορετικά απλά χάνουμε το χρόνο μας και εξαπατούμε τον κόσμο. Και εγώ πρώτα απ' όλους δεν θέλω να εξαπατήσω κανέναν και ούτε θέλω κι εγώ να με κοροϊδεύουν. Είναι ένα θέμα πολύ λεπτό, για το οποίο γίνεται πολλής λόγος, αλλά δεν γίνονται στην πράξη πολλά πράγματα. Επιθυμούν οι συνάδελφοι να λάβουν τον λόγο. Όχι, εσείς κυρία μου τότε. Η κυρία Τζερομέτα είναι η αναφέρουσα. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση σε σχέση με τα όσα είπε ο εκπρόσωπος της κυβερνήσης μας. Εκείνος μίλησε για τραπέζια. Τραπέζια συζήτηση. Αυτά γίνανε πριν από τρία χρόνια. Ούτε ένα διάταγμα δεν έχει εκδοθεί. Έχουμε επίγον πρόβλημα που αφορά την υγεία του κόσμου. Και πιστεύουμε ότι η κυβέρνησή μας μπορεί και οφείλει να κάνει πολλά περισσότερα τώρα να δώσει απόλυτη προτεραιότητα σε κάθε επίπεδο, περιφερειακό, τοπικό, εθνικό, στο πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Η Ιταλία έχει τον μεγαλύτερο αριθμό πρώιμων θανάτων στην Ευρώπη, με, ανάμεσα σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και θα ήθελα να πω ότι μόλις βλέπω εδώ έκδοση τον Απρίλιο του 2016 ένα έγγραφο από τη Γενική Διεύθυνση για Εσωτερική Πολιτική του Ευρωκοινοβουλίου που μιλά συγκεκριμένα για την κατάσταση του Μιλάνο και μάλιστα σε αυτό το έγγραφο επιβεβαιώνεται ότι μπλοκάριστηκαν και αφαιρέθηκαν μέτρα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να πιέσουμε τις περιφερειακές και την εθνική μας κυβέρνηση ώστε να μπορούν και να δραστηριοποιηθούν με τις πολιτικές τους. Εγώ αντιπροσωπεύω μία ένωση που ονομάζεται Πολίτες για τον Αέρα. Ε, πριν από λίγες μέρες στείλαμε επιστολή στον Πρωθυπουργό Ρέντζη ζητώντας μεγαλύτερη δέσμευση και συμμετοχή για την οδηγία ΝΕΚ γιατί είναι προφανές ότι πρόκειται για πολιτικές αλληλένδετες. Ε, δεν μπορεί δηλαδή να μιλάμε, δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα για παράδειγμα των ε, δοκιμών ε, σε πραγματικές ε, συνθήκες οδήγησης χωρίς να μιλάμε για το θέμα της υγείας και του αέρα. Αυτό κάνει όμως η κυβέρνησή μας. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα αλλάξει η τακτική. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται για ένα υπαρκτό πρόβλημα. Μα ικανοποιεί το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτελεί το καθήκον της, αναμένουμε τις πληροφορίες που θα μα χορηγήσει προσεχώς και αναμένουμε να επικοινωνήσει και με την Ιταλική κυβέρνηση. Αν συμφωνείτε όλε και όλοι θα μείνει ανοιχτή η αναφορά μέχρι ότου λάβουμε νεότερες πληροφορίες. Ακολουθεί το υπαριθμόν 14 αναφορά του κ. Μάης, Βέργου σχετικά με την ρήπανση στην Αμβέρσα. Πρόκειται για την κυρία μας, συγγνώμη. Εδώ είμαι, με συγχωρείτε. Κύριε Πρόεδρε, μέλη της Κοινοβουλευτικής Αυτής Επιτροπής, όλοι παρόντες, υπέβαλα την αναφορά μου τον Νοέμβριο του 2011, ανησυχώντας για την ποιότητα ζωής στην Αβέρσα. και ιδιαίτερα ανησυχώντας για την υγεία των κατοίκων της. Ακόμα και οι γιατροί κρούν συνεχώς τον κόδωνα του κινδύνου εξαιτία της μεγάλης συχνότητας λοιμόξεων των αναπνευστικών οδών στα παιδιά της πόλης μας. Για να εξηγήσω. Η Αμβέρσα είναι μια πόλη η οποία έχει γύρω της τέσσερις μεγάλους δακτυλίους και επιπλέον γύρω από αυτού υπάρχουν και αυτοκινητόδρομοι που οδηγούν στη Γάνδη, στις Βρυξέλλες, μέσα από το Μπομ και μέσα από το Μάχελεν, στη Λιέγη, στο Εντχόβεν, στο Μπέργεν και στο Ζόμ και στην Πρέντα. Το κυκλοφορικό είναι τεράστιο. Οι είναι καθημερινά μεγάλες, όλο και περισσότερες. Μέρα και νύχτα χρησιμοποιούνται εντατικά οι δρόμοι μας. Αυτό όμως που με απασχολεί εμένα είναι ότι παίρνονται όλο και περισσότερα μέτρα στην Αβέρσα ώστε το δικό δίκτυο να χρησιμοποιείται όλο και πιο εντατικά. Και τι εννοώ, ότι μεγαλώνει το λιμάνι, πράγμα που σημαίνει ότι και το κυκλοφοριακό λίγο από το λιμάνι μεγαλώνει, μεγαλώνει το αεροδρόμιο τη Αβέρσα, όπου πια πηγαίνουν και τακτικέ πτήσει και καταλαβαίνω ότι όλα αυτά γίνονται στο όνομα τη οικονομία. Αλλά η οικονομία πρέπει να φροντίσει να υπάρχει και μια καλή ρύθμιση για την κοινωνία και στη βάση κάθε καλή οικονομία τελικά είναι οι υγιείς άνθρωποι, υγιείς ε, εργαζόμενοι και επιχειρηματίες. Δεν λέω ότι μόνο το κυκλοφοριακό φταίει για την κατάσταση, αλλά σίγουρα δεν είναι και αθώο. Το Βέλγιο πολλές φορές έχει κληθεί να απολογηθεί για την παραβίαση της οδηγίας όσον αφορά την ποιότητα του αέρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πράγματι, είναι γεγονός ότι στην Αβέρσα το λιμάνι της τα τελευταία 30 χρόνια έχει αυξηθεί όσον αφορά την δυναμικότητά του με πάνω από 50% τα τελευταία 15 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ενώ το 1985 είχαμε 80 εκατομμύρια, το 2000 είχαμε πάνω από 120 και πάνω από 200 εκατομμύρια τόνους το 2015. Αυτό σημαίνει ότι αν συνεχίσουμε με αυτό το αριθμό το 2030 η χωρητικότητα θα είναι πάνω από 300 εκατομμύρια τόνοι. Και όλα αυτά τα εμπορεύματα, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να μεταφερθούν με τις μεταφορές, ε, οδικό σε ένα μεγάλο βαθμό. Και παρόλο που είχαν πει ότι ποσοστία θα φροντίσουν να μειωθούν οι οδικές μεταφορές κατά 56% για την απομάκρυνση των εμπορευμάτων αυτών, τελικά παρόλα αυτό υπάρχει αύξηση 50%. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι για να δοθεί περισσότερος χώρος στους δρόμους κόβονται δέντρα, μειώνονται πράσινοι χώροι, το δάσος της ε, Αγίας Άννας, για παράδειγμα, το Νόρτ Καστέλ, αλλά ακόμα και μικρές πλατείες με πράσινο καταργούνται. Πολλές λοιπόν οργανώσεις πολιτών στην Αβέρσα διαμαρτύρονται. Υπάρχει οργάνωση Ρίγκλαντ, η οποία ζητάει να καλυφθεί το ring, ο δακτύλιος δηλαδή, να σκεπαστεί. Υπάρχει οργάνωση Straten General, που και αυτή ζητάει η σύνδεση με το ποτάμι Σχέλντε να γίνει εκτός της πόλης αλλά και διάφορε τοπικέ ομάδες κατοίκων επίσης δραστηριοποιούνται για να μην κόβονται τα δέντρα στι γειτονιές τους. Πρέπει να δούμε ότι τελικά στην Αβέρσα όλοι ζούμε μέσα στην κυκλοφορία. Ακόμα και τα σχολιά βρίσκονται δίπλα σε αυτοκινητόδρομους. Διαπιστώνω επίσης ότι με αδιαφορία αντιμετωπίζονται οι ελεύθεροι χώροι. Γιατί αυτό που γίνεται είναι ότι και αυτοί κτίζονται τελικά. Στον Πέρχεμο που εγώ ζω έχει χτιστεί μια μεγάλη πολυκατοικία με γραφεία που σημαίνει λιγότερα δέντρα και περισσότερη κυκλοφορία. Είναι το CityLink. Για να μην είμαι όμως μόνο αρνητική για όλα αυτά, πρέπει εδώ να σημειώσω ότι γίνονται έρευνες για την ποιότητα του αέρα στην Αβέρσα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που ονομάζεται κυρίως Ζενέζο, περίεργες μύτες δηλαδή, που ακριβώ εξετάζει την ποιότητα του αέρα που κοινού με πανεπιστήμια. Επίση, το γεγονό ότι προσφέρονται περισσότεροι ποδηλατόδρομοι και αυτό είναι θετικό. Και δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μέτρα για την κυκλοφορία. Αυτό που, που με ενδιαφέρει είναι η υγεία του κόσμου. Γιατί και αυτή η υγεία είναι μια πτυχή της οικονομίας. Το επιχείρημά μου λοιπόν ήταν και παραμένει ότι περισσότερος χώρος για τις οδικές μεταφορές εμποδίζει την δουλειά που θα έπρεπε να γίνει για εναλλακτικέ λύσεις, για την αποκέντρωση, για το να δουλεύουμε από το σπίτι, για να μετακινούμαστε μόνο όταν είναι πραγματικά ανάγκη. Με δύο λόγια, εγώ θα ήθελα να μην καταλήξει η Αβέρσα ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος, αλλά να παραμείνει ένας χώρος που να μας αρέσει να ζούμε, να εργαζόμαστε και να υποδεχόμαστε τους φίλους μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέρω ότι ο δικό σα ρόλο είναι να αποφασίσετε για το στόχο και όχι για τα μέσα. Οπότε ίσω οι πολίτε είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να φροντίσουν να γίνει έρευνα και να αποφασίζουν βάσει αποτελεσμάτων. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. Παρακαλώ την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ενημερώσω την απάντηση που έχει δώσει ήδη από το Δεκέμβριο του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τότε είχαμε στη διάθεσή μας δεδομένα του 2014. Τα δεδομένα του 2015 ακόμη δεν είναι διαθέσιμα και δεν μπορώ να κάνω τη σχετική ενημέρωση. Μπορώ όμως να σας πω τι γίνεται με την διαδικασία προσφυγής. Στην απάντησή μας αναφέρουμε ότι θα προσφύγουμε κατά του Βελγίου διότι δεν τηρεί τις οριακές τιμές των PM10. Εδώ τώρα η κατάσταση είναι σήμερα λίγο διαφορετική διότι δεν έχει εκτελέσει την απόφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσφύγει στο δικαστήριο. Όταν έλαβε την απόφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι διαθέσιμες πληροφορίες ήταν για το έτος αναφοράς 2013 και μας έδειχναν ότι το Βέλγιο δεν είχε σεβαστεί τις οριακές τιμές PM10 για αστικές περιοχές. Το 2014 η κατάσταση άλλαξε. Οι, αναφο οι ποιότητας έδειξαν ότι το Βέλγιο είχε τροποποιήσει τη στάση του σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Βρυξέλλες, Γάνδη, η ε, περιφέρειες των λιμανιών και κέντρα άνω, κέντρα άνω των 50.000 κατοίκων. Έχει αλλάξει λοιπόν η κατάσταση σήμερα. Η ΔΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή απεφάσισε να αναστείλει την απόφαση αυτή για την προσφυγή κατά του Βελγίου. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανεξετάσει την κατάσταση όταν θα είναι διαθέσιμα τα δεδομένα για το έτος 2015. Αυτό θα συμβεί τον Σεπτέμβριο του 2016. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Βέλγιο τηρεί όλες τις οριακές τιμές των PM10, διότι υπάρχει μία ε, ζώνη η οποία δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις οριακές τιμές, η οποία όμως δεν είχε περιληφθεί στην αρχική προσφυγή. Γιατί την εποχή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ανοίξει την διαδικασία προσφυγής, η περιφέρεια αυτή ήταν, βρισκόταν εντός των πλαισίων των ενεργειακών τιμών. Έτσι δεν περιλήφθηκε λοιπόν στην αρχική προσφυγή λόγω παραβίασης. Όλες οι άλλες ζώνες, ωστόσο, συμμορφώνονται τώρα, σύμφωνα με τα δεδομένα του 2014. Θα επανεξετάσει λοιπόν, όπως εξήγησα, την κατάσταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν, τον Σεπτέμβριο 2016, θα έχουμε στη διάθεσή μα τα δεδομένα του 2015. Θα αποφασίσουμε τότε για τα επόμενα βήματα που θα λάβουμε και για το εάν θα προσφύγουμε στο δικαστήριο κατά του Βελγίου για υπέρβαση των οριακών τυπών. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Ο κύριος Μπαρτ Στάς είναι εδώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Μάσεν, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαι μέλος της Επιτροπής αυτής, της Κοινοβουλευτικής, αλλά και της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, παρακολουθώ πολύ τι γίνεται όσον αφορά την ποιότητα του αέρος. Οπότε, Γνωρίζω την κατάσταση στην, Αβόρ, στην Αβέρσα. Την κυρία Μες πρέπει να ομολογήσω ότι δεν την είχα γνωρίσει προσωπικά μέχρι πρόσφατα. Μόνο με την πρωτοβουλία της αυτή στην κοινοβουλευτική διαδικασία τη γνώρισα. Και πρέπει να πω ότι οι απαιτήσει της, η επιχειρηματολογία της είναι κάτι που αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά και στηρίζω. Η Επιτροπή τώρα μας λέει ότι τα νούμερα, τα οποία είναι γνωστά, έχουν κάποιες αλλαγές κατά πάσα πιθανότητα με αυτά του Σεπτεμβρίου του 2016, οπότε θα παρακολουθεί την κατάσταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, προφανώς, φυσικά, ανάμεσα από το 2012 και με το 2015, όμως ξέρουμε τι έχει γίνει, οπότε μακάρι να αλλάξει κάτι. Πολύ θα χαρούμε. Όμως το θέμα της ποιότητας του αέρα είναι πάρα πολύ σοβαρό στην περίπτωση της Αβέρσας και έχει τεράστιες επιπτώσεις στη ζωή και τη δουλειά των ε, κατοίκων της πόλης αυτής και κυρίως επηρεάζει την υγεία των παιδιών. Η κυρία Μάση μας ε, το είπε ότι πάρα πολλά σχολεία έχουν καταλήξει να βρίσκονται δίπλα σε αυτοκινητοδρόμους. Το ρίγκο δακτήλιος που δεν είναι ουσιαστικά δακτύλιο στην αβέρσα γιατί περνάει μέσα από, την πόρτα, από το κέντρο της πόλης. Οπότε και δημοτικά και γυμνάσια αλλά και παιδικοί σταθμοί ακόμα βρίσκονται κοντά σε αυτούς. Καταλαβαίνετε ότι η υγεία των παιδιών μας κινδυνεύει. Δεν είναι μόνη της η κυρία Μάσεν. Αυτή δεν είναι αναφορά ενός μεμονωμένου ατόμου. Η κυρία Μάσεν μας είπε ότι εκφράζει το αίσθημα όλων των κατοίκων της Αβέρσας. Υπάρχουν διάφορες επιτροπές δράσης πολιτών. Η μία είναι η Straten General, η άλλη είναι το Αντεμλός, δεν μπορώ να αναπνεύσω σημαίνει Αντεμλός. Είναι και αυτή μια επιτροπή δράσης που ακριβώς ασχολείται με το θέμα της ρήπανσης του αέρα. Υπάρχει Ringland, είναι μια επιτροπή αυτή η οποία εξετάζει το θέμα του αυτοκινητόδρομου, όπου και εκεί υπάρχουν προβλήματα με την ποιότητα του αέρα. Και πριν από μερικά χρόνια υπήρξε ένα δημοψήφισμα. Οργανώθηκε από τις οργανώσεις αυτές. Σήμερα το πρωί πρέπει να σας πω ότι από ό,τι φαίνεται η τοπική κυβέρνηση αλλά και η φλαμανδική και η περιφερειακή κυβέρνηση φαίνεται ότι σιγά σιγά έχοντας μιλήσει μεταξύ τους καταφέρνουν να ακούνε ο ένας τον άλλον. Η κυρία μας μας είπε ότι υπάρχει και ένα σχέδιο, το κυρίως Ζενέζεν, που είναι ένα επιστημονικό πρόγραμμα, όπου 2.000 κάτοικοι γνωρίζουν, ε, επιστημονικά θέλουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, βάζοντας ε, σε διάφορα σημεία, σε πολλές γειτονιές της πόλης, αλλά και κυρίως για να ευαισθητοποιήσουν περισσότερο τον κόσμο. Άκουσα την απάντηση της Επιτροπής. Αυτή που μόλις ακούσαμε, ότι περιμένουν τις καινούργιες πληροφορίες. Με τις πληροφορίες που έχουμε στο φάκελό μας. Πιστεύω ότι, η αναφορά αυτή πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και η δράση της κυρίας μας να ληφθεί υπόψη. Γι' αυτό λοιπόν, Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας ζητήσω να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή. Μετά από τόσα μας είπε η κυρία μας, για να παρακολουθήσουμε το τι γίνεται στην Αβέρσα, πώς θα προχωρήσει αυτή η υπόθεση, ώστε στην πόλη να υπάρχει ένα καλό κλίμα, μια καλή ατμόσφαιρα, οι άνθρωποι να ζουν καλά, να μην κινδυνεύει για τον κατοίκον της, ούτε και οι τουρίστες που είναι πολύ άριθμοι και μας επισκέπτονται εκεί. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Άλλος κανείς θέλει το λόγο παρακαλώ για αυτή την αναφορά. Α, τότε κυρία μας. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας έτσι κι αλλιώς το χώρο που παίρνουν οι δρόμοι. Δεν έχει να κάνει αυτό μόνο με την οδηγία. την ε, Αμβέρσα δεν υπάρχει καμιά γειτονιά από την οποία να μην περνάει ένας αυτοκινητόδρομος. Ζητάω λοιπόν αυτήν την ιδιαίτερη προβληματική να τη λάβετε υπόψη σας. Έπειτα, με τους πολίτες που έχω μιλήσει εγώ, σκέφτομαι ότι αυτονό την επιθυμία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Αυτοί διαμαρτύρονται. Υπάρχει τεράστια ανησυχία από τους πολίτες της Ανβέρσας εξαιτίας του γεγονότος ότι το κυκλοφοριακό αυξάνεται συνεχώς. Τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Η κατάσταση είναι αφόρητη. Στην Αβέρσα δεν βλέπετε τίποτα άλλο παρά από δύο λουρίδες με φορτηγά. Ο κύριος Στάς ζήτησε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή. Και αν καταλαβαίνω καλά και από τους άλλους αναφέροντες, είναι ένα πρόβλημα αυτό της ρήπανση στο αέρος που είναι σε ολόκληρη την Ευρώπη ένα πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι έχετε δίκιο. Βλέπουμε και εμείς ότι πρόκειται για μεγάλο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη λαμβάνουμε πολλές σχετικές αναφορές. Η αναφορά σας θα παραμείνει ανοιχτή. Θα περιμένουμε τις απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο. Η Κομισιόν θα συνεχίσει τον διάλογο με την βελγική κυβέρνηση και θα επανέλθουμε. Ο κύριος Πέτερ Γιάρ. Σωστά το είπατε. Η Κομισιόν είπε ότι θα λάβουμε απάντηση τον Σεπτέμβριο και ας σημειώσουμε κι εμείς να επανέλθουμε τον Σεπτέμβριο να μάθουμε εάν έχει υπάρξει κάποια ε, καινούρια απάντηση ή εν πάση περιπτώσει να επανέλθουμε στο θέμα ε, το φθινόπωρο. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, μπορούμε να προχωρήσουμε στο τελευταίο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Πρόκειται για 13 αναφορές σχετικά με μια εγκατάσταση στον βιομηχανικό λιμένα στη Λάρνακα. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Έντιμε κύριε Πρόεδρε, έντιμα μέλη. Βρίσκομαι εδώ σήμερα εκπροσωπώντας τους πολίτες της Λάρνακας για να σας παρουσιάσω την κατάσταση στο λιμάνι της πόλης μας, μιας όμορφης παραθαλάσσιας πόλης της Κύπρου. Δυστυχώς, τον Ιούνιο του 2014, στο λιμάνι της πόλης μας εγκαταστάθηκαν μονάδες βαριάς βιομηχανίας, οι εργασίες των οποίων συνδέονται με την εξόριξη ανθράκων στην Κυπριακή ΑΟΣ. Έκτοτε, εκατοντάδες κάτοικοι διαμαρτυρόμαστε έντονα, εφόσον το λιμάνι βρίσκεται εντός του αστικού ιστού της Λάρνακας, σε απόσταση μόλις μερικών μέτρων από σπίτια και δίπλα από τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη παραλία λουμένων της πόλης, τη διάσημη παραλία των Φινικούδων, όπου κολυμπούν χιλιάδες τουρίστες, αλλά εμείς και τα παιδιά μας. Το λιμάνι της Λάρνακας είναι ένα μικρό σε έκταση λιμάνι, τοποθετημένο στο κέντρο της πόλης, μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Πρόκειται για το δεύτερο σε μέγεθος λιμάνι της Κύπρου και είναι εμπορικής και τουριστικής χρήσης. Τον Ιούνιο του 2014 πληροφορηθήκαμε από ανεπίσημες πηγές ότι στο λιμάνι μας θα εγκαθίσταντο δύο οχληρές μονάδες προς εξυπηρέτηση των εταιριών υδρογονανθράκων. Οι συγκεκριμένες οχληρές εγκαταστάσεις αποτελούνται από μονάδα παραγωγής υγρής λάσπης, liquid mud plant, και αποθήκη χημικών σε απόσταση μόνο 125 μέτρων από σπίτια. Να σας ενημερώσω επίσης ότι επί καθημερινής βάσεως θα γίνεται διακίνηση βαρέων οχημάτων εντό των κύριων οδικών αρτηριών τη πόλη, μέσα από κατοικημένε περιοχέ προ δύο εργοστάσια υποστηρίξη των εταιριών Χάλιμπαρτον και Σλάμπερκερ, τα οποία και πάλι έχουν παράτυπα ανεγερθεί εντό μια ζώνη ελαφριά βιομηχανία, ενώ πρόκειται για μονάδε βαριά βιομηχανία και τα οποία βρίσκονται σε απόσταση μόλι 800 μέτρων από τα πλησιέστερα σπίτια. Οι κυβερνητικέ αποφάσει για εγκατάσταση των εν μονάδων στο λιμάνι Λάρνακα κρίνουμε ότι παραβιάζουν τα ακόλουθα. Τη σύμβαση του Άρχου, την οδηγία 96 κάθετο 82, την οδηγία 2012 κάθετο 18, 2003 κάθετο 4, 2001 κάθετο 41. Να αναφέρω ότι ω κάτοικοι δεν είχαμε έγκαιρα όπως προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία την αναγκαία πληροφόρηση και δεν λάβαμε ποτέ επίσημη πληροφόρηση αναφορικά με το είδος και τις ποσότητες χημικών ουσιών που αποθηκεύονται στις συγκεκριμένες μονάδες. Δεν πληροφορηθήκαμε με ποιο ακριβώς τρόπο γίνεται η διαχείρισή τους, ούτε ποια μέτρα έχουν ληφθεί προς αποτροπή ατυχήματος, ανάφλεξης ή έκρηξης. Επίση δεν μας ενημέρωσαν με ποιο τρόπο θα πρέπει να αντιδράσουμε σε περίπτωση ατυχήματος δεν λάβαμε ποτέ μέρος στον καταρτισμό εξωτερικών σχεδίων επίγουσας ανάγκης, ως προσβλέπεται από το άρθρο 8 της Οδηγίας 96 82. Δεν υπήρξε καμία ενημέρωση του κοινού για τη συμμόρφωση ή μη της κυβέρνησης με την υποχρέωση που πηγάζει από το άρθρο 9 της Οδηγίας 96-82. Τέλος, αλλά πάρα πολύ σημαντικό, κρίνουμε ότι έχουν παραβιαστεί διατάξεις της Οδηγίας 2001 42 σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων στο περιβάλλον λόγω του κινδύνου ατυχημάτων και συνακόλουθα των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Καταληκτικά σχόλια. Η χρήση του λιμανιού Λάρνακα ω εφοδιαστική βάση για την εξυπηρέτηση εταιριών υδρογονανθράκων, αλλιώ βάση logistics, εμπεριέχει κινδύνου για το περιβάλλον λόγω του ενδεχομένου πρόκληση ατυχήματο συνακόλουθα δε για την ασφάλεια και υγεία των κατοίκων. Επιπρόσθετα, η εφοδιαστική βάση εξαρτάται από βιομηχανικές περιοχές, στις οποίες εγκαθίστανται άλλες υποστηρικτικές εταιρείε για την εξυπηρέτηση της βιομηχανίας συντρογών ανθράκων. Αυτές οι περιοχές βρίσκονται πολύ μακριά από το λιμάνι της Λάρνακας, κάτι το οποίο αναγκάζει τα οποιαδήποτε φορτία με κρυκτικά, ραδιενεργές πηγές, απόβλητα και σωλήνες που ενδεχομένω να περιέχουν ραδιενεργά στοιχεία, να διακινούνται διαμέσου της πόλης, περνώντας μπροστά από σπίτια και σχολεία, όπου αυξάνεται ο κίνδυνος ενδεχομένου ατυχήματος με επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην υγεία και ασφάλεια των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και ευελπιστώ ότι η απόφασή σας κατά τη σημερινή εξέδαση του σημαντικού αυτού θέματος, το οποίο επηρεάζει τις ζωές χιλιάδων πολιτών και το μέλλον μιας πόλης, θα διασφαλίσει την υγεία και ασφάλειά μας και θα υποχρεώσει το κράτος να ακολουθήσει τις νενομισμένες διαδικασίες. Και τέλος, θα ήθελα να καλέσω την Επιτροπή, όπως έρθει στη Λάνακα, για να δει επιτόπου το πρόβλημά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Eh, ευχαριστώ πολύ. Η εκπρόσωπος της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαριστεί την Επιτροπή Αναφορών που μας προσφέρει την ευκαιρία να προσέλθουμε να της απευθύνουμε τον λόγο καθώς και στις αναφερόμενες και αναφερόμενους. Θα ήθελα πρώτα να σημειώσω ότι υπάρχουν καταγγελίες που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό Έχουν υποβάλει και πολλές σχετικές πληροφορίες οι καταγγέλλοντες. Η Κομισιόν έχει απαντήσει σε έναν αριθμό αναφορών που εξετάζονται και εδώ ήδη από τον Νοέμβριο του 2015. Νομίζω ότι από τότε δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Θα ήθελα να σημειώσω αναφορικά με την Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία, τις οποίες ε, οδηγίες θύμισε η αναφερομένη. Πρώτον, όσον αφορά τη συνθήκη άρχους, οι απαιτήσει της έχουν περιληφθεί σε επιμέρους ειδικέ περιβαλλοντικές οδηγίες. Περιλαμβάνονται λοιπόν στην ε, εκάστοτε οδηγία. Πρώτα λοιπόν σε ό,τι αφορά την οδηγία που αποκαλείται οδηγία Σεβέζο 9682 και την οδηγία 2012-18. Σημειώνω ότι η δεύτερη δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή, διότι άρχισε να ισχύει από 1η Ιουνίου 2015. η ΔΕ Οδηγία 9682, οφείλω να σημειώσω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμπεραίνεται ότι οι εγκαταστάσεις αυτές εμπίπτουν σε αυτή την οδηγία, διότι οι ουσίες και ποσότητες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αυτής. Το μόνο θέμα έχει να κάνει με την χωροταξία, με το χωροτακτικό σχεδιασμό δηλαδή. Επειδή αναγνωρίζεται, υπάρχουν αναγνωρισμένες εγκαταστάσεις σε βέζο μέσα στο λιμάνι, έχουμε, ή μάλλον δεν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι κυπριακές αρχές δεν έχουν εφαρμόσει ή πάντως δεν έχουν ορθώς αξιολογήσει τις αποστάσεις των υφισταμένων εγκαταστάσεων από τις νέες και τώρα σε ό,τι αφορά την 141-2001 SEA ούτε αυτή εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή διότι αυτή αναφέρεται σε εγκαταστάσεις και προγράμματα και όχι σε έργα, project δηλαδή όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση όπου εδώ εφαρμόζεται η οδηγία περιβαλλοντικού αντικτύπου. Τα έργα δε αυτά εμπίπτουν στο παράρτημα 2 της σχετικής οδηγίας, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει υποχρέωση της χώρας μέλους να διεξαγάγει μελέτη επιπτώσεων, παρά μόνο προκαταρκτικού screening που από τις πληροφορίες που έχουμε λάβει αυτό έχει γίνει. Στην δε περίπτωση αυτή, η χώρα μέλος υποχρεούται μόνο να ενημερώσει το κοινό, δεν υποχρεούται να προβεί σε διαβούλευση. Ωστόσο, από όσα αντιλαμβανόμαστε, τον Ιούλιο του 2014 έγινε μια information session ανοιχτή στο κοινό, που ακολουθήθηκε και από δύο συναντήσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών, όπου το κοινό μπορούσε να συμμετάσχει και για τον λόγο αυτό, στην υπόθεση αυτή δεν μπορεί να συμπεράνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρόκειται για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον από τις προφορίες που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει ως τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. συνάδελφοι, ο κύριος Παπαδάκης. Είναι προφανές ότι υπάρχει διάσταση μεταξύ των ε, παραπονούμενων πολιτών και της απάντησης που λάβαμε μόλις τώρα από την Επιτροπή. Θεωρώ ότι δεν έγιναν οι απαραίτητες διαδικασίες, ούτε οι ορθές περιβαλλοντικές μελέτες για αυτό το συγκεκριμένο ζητούμε θέμα, αλλά ούτε και ο δημόσιος διάλογος είτε ενημέρωση όπως ελέγχθη προλίγου. Γι' αυτόν πιστεύω ότι το θέμα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό. Ταυτόχρονα ε, να και πολύ αυστηρές συστάσεις προς την Κυπριακή Δημοκρατία για την εφαρμογή όλων των απαρατητουμένων απαραίτητων διαδικασιών όπου πρέπει να ακολουθούνται πιστά για τους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σάλφε. Ευχαριστώ. Εσείς ο κύριος Νομίζω ότι τα θέματα περιβάλλοντος και αναφέρομαι βεβαίως και στο συγκεκριμένο θέμα που έχουμε μπροστά μα υπό συζήτηση αλλά και γενικότερα αναφερόμενοι σε θέματα περιβάλλοντος πρέπει να αναχθεί και είναι κυρίως υποχρέωση των εκπροσώπων των πολιτών των ευρωπαϊκών λαών να το ανάγουν σε μέγιστη σημασία ζήτημα όχι μόνο γιατί επηρεάζει την υγεία των πολιτών αυτής της Υπήρου αλλά γιατί το περιβάλλον αποτελεί, θα πρέπει να αποτελεί μέσα στο μυαλό μας το μεγαλύτερο ζήτημα που έχει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα για την επιβίωση του πλανήτη. Κάτω από αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να διευρυνθεί η οπτική με την οποία αντιμετωπίζουμε ζητήματα που καταγγέλουν οι πολίτες γιατί η αυστηρή προσήλωση στο τι λένε οι οδηγίες τις οποίες ασφαλώς πρέπει να ακολουθούμε συνεπάγεται κατά τη δική μου κρίση ότι μειώνομαι την αντίληψη, το μέγεθος της αντίληψης που έχουμε για το τι σημαίνει περιβάλλον στον σύγχρονο κόσμο. Και δεν θα το διευρύνω περισσότερο, διότι μιλώ σε ανθρώπους που έχουν πολύ στενή σχέση με τα θέματα περιβάλλοντος. Η αναφορά της εκπροσώπου της ε, Επιτροπής εδώ ότι υπάρχει οδηγία η οποία είναι μεταγενέστερη της καταγγελίας, τουλάχιστον έτσι το έχω καταλάβει, ε, και θα χρειαστώ ίσως μια διευκρίνηση, ε, νομίζω ότι τη δική μου νοημοσύνη την βάζει σε ένα προβληματισμό. Επίσης έχει λεχθεί ότι δεν υπάρχει παραβίαση των περιβαλλοντικών κανόνων και κατέληξε η εκπρόσωπος της Επιτροπής σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες. Αλλά δεν γνωρίζω πόθεν ήρθαν αυτές οι πληροφορίες, αν είναι μόνο από την κυβερνητική πλευρά ή αν υπάρχουν έρευνες περι... περιβαλλοντικής μελέτης οι οποίες έχουν ε, ληφθεί ή δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Η, προσπάθεια για δημιουργία ε, τέτοιου εργοστασίου ουσιαστικά τοξικών ουσιών σε ένα χώρο που γυπνιάζει ε, κατοικιών, σε μια πόλη η οποία υποφέρει ήδη από τους ρήπους είτε των αποθηκών καυσίμων που είναι στην περιοχή εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, είτε και του αεροδρομίου προσθέτοντας εδώ ότι και οι δύο αυτές εγκαταστάσεις ε, είναι παραθαλάσσιες σε μια τουριστική πόλη. Το γεγονός επίσης ότι ε, οι ήδη οι κάτοικοι έχουν καταγγείλει ότι δεν υπήρξε ενημέρωση και διαβούλευση με την κυβέρνηση αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρνακας ε, αντέδρασε απέναντι σε αυτή την ε, κυβερνητική απόφαση. Και νομίζω σωστό εδώ να υπομνήσουμε ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ε, κατεξοχήν εκπροσωπούν ε, τους πολίτες της πόλης. Θεωρώ ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει τουλάχιστον, για να μην πω κάτι πιο συγκεκριμένο, πιο ηχηρό, να κρατήσει αυτό το θέμα στην ατζέντα της και να ξαναζητήσει, να ζητήσει τις ε, αναγκαίες διευκρινήσεις για το αν υπάρχουν ε, οι αναγκαίες περιβαλλοντικές μελέτες και να γνωρίζει ο πολίτης της πόλης ότι αυτές οι, αυτές μελέτες έχουν καταδείξει αυτό ή το άλλο. Αυτή η υπόθεση θα πρέπει να απασχολήσει ξανά την Επιτροπή μας και ε, υπογραμμίζω και εγώ ότι μια επίσκεψη στην περιοχή όπως έχει ήδη αναφέρει εδώ η αναφέρουσα το θέμα ε, συμπολίτισμου. Ε, μια επίσκεψη λοιπόν στην περιοχή νομίζω ότι ε, θα κρίνει πάρα πολλά για το μέλλον αυτής της υπόθεσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μαριά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε σημαντικές ε, αναφορές οι οποίες ε, έχουν σχέση με το θέμα και φυσικά μία εκπρόσωπο η οποία όμως μας ενημέρωσε για όλες τις αναφορές και θα έλεγα με ένα πολύ σαφή τρόπο. Προκύπτει λοιπόν εδώ ότι αυτή η προσπάθεια στην Κύπρο για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων ε, αρχίζει και δημιουργεί προβλήματα. Και αν η Κύπρος θέλει πράγματι να γίνει ένα κέντρο σοβαρό όπου θα έχουμε εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Θα πρέπει να υπάρξει ένα συνολικό σχέδιο, ούτως ώστε με την ανάπτυξη ε, πράγματι της έρευνας για τους υδρογονάνθρακες και να μην δημιουργούνται προβλήματα στο περιβάλλον και να μην κινδυνεύει, κινδυνεύουν άλλοι τομείς της οικονομίας όπως είναι τα θέματα του τουρισμού, της αλληλείας και γενικότερα οικονομικές δραστηριότητες και φυσικά να μπει μέσα σε ένα σχέδιο. Και τέτοιο σχέδιο δεν έχουμε δει, διότι βλέπουμε ξαφνικά εγκατάσταση αυτών των δραστηριοτήτων, βλέπουμε δραστηριότητες που γίνονται σχεδόν στα όρια της πόλης, σε μικρή απόσταση, βλέπουμε ένα λιμάνι το οποίο μπορεί να ήταν και επιβατικό και να έχει και άλλες χρήσεις ξαφνικά να μπλοκάρεται από αυτές τις διαδικασίες που οι συγκεκριμένες εταιρείες ε, θέλουν να κάνουν λόγω των, της αξιοποίησης των ανθράκων Επομένως, έχουμε ένα σοβαρό θέμα και δεν είναι μόνο στο παρελθόν τι γίνεται, αλλά είναι και στο μέλλον. Το δεύτερο θέμα, αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπε η Επιτροπή, εγώ κατάλαβα ότι υπάρχει παραβίαση της οδηγίας που ονομάζεται οδηγίες Σοβέζο. Εγώ αυτό κατάλαβα. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει να μας πει υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις θα προχωρήσει στον έλεγχο αυτής της παραβίασης των ε, οδηγιών, εκτός αν υπήρχε πρόβλημα στη Δερμηνία. Εγώ έτσι άκουσα να λέει η Επιτροπή. Δεύτερον, το γεγονός ότι έχουμε οδηγίες που ισχύουν μεταγενέστερα δεν σημαίνει ότι δεν υφίσταται παραβίαση, διότι οι παραβιάσεις σε σχέση με τα περιβαλλοντικά είναι συνεχείς και υπάρχουν. Επομένως και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας ε, απασχολήσει. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα εργοστάσιο τοξικών στην ουσία, το οποίο απέφχομαι να δημιουργήσει πολύ σοβαρό πρόβλημα στο μέλλον. Έχουμε προβλήματα δημόσιας υγείας και νομίζω ότι πρέπει κανείς να τα δει πολύ πιο σοβαρά. Επομένως, πρώτον, θα πρέπει κατά την άποψή μας, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, να κρατηθεί ανοιχτή η συγκεκριμένη αναφορά. Δεύτερον, να γίνει επιστολή στο Δήμο της ε, Λάνακας εν προκειμένου για να τοποθετηθούν, διότι δεν έχουμε μια ενημέρωση από τον ίδιο το Δήμο πώς βλέπει το θέμα και πώς σκέπτεται να το αντιμετωπίσει. Το τρίτο είναι προφανές ότι πρέπει να στείλουμε επιστολή στις κυπριακές αρχές, ούτω ώστε να εκφράσουμε την ανησυχία μας, να εκφράσουμε τον προβληματισμό μας και να μας πούν πώς προβλέπουν να αντιμετωπίσουν στο μέλλον αυτό το ζήτημα. Και επιμένω, εφόσον η Κύπρος στρατηγικά μπαίνει σε μια λειτουργία αξιοποίησης των υδρογονανθράκων, δεν μου φαίνεται σοβαρή η στρατηγική που προετοιμάζεται για να αξιοποιήσει αυτή τη διαδικασία. Είναι δύο πλατφόρμες που βρίσκονται στη θάλασσα σε απόσταση 8 χιλιόμετρων από το σημείο, από τη Λάρνακα και από το σημείο που συζητούμε και αν ξαφνικά για τις δύο πλατφόρμες έχει δημιουργηθεί αυτή η κατάληψη του χώρου του, ε, του λιμανιού και όλα αυτά τα προβλήματα, τι θα γίνει αν Κύπρος αναπτύξει σοβαρά όλη την βιομηχανία ας πούμε αξιοποίησης και άντλησης υδρογονανθράκων. Τι θα γίνει το νησί. Επομένω είναι ευκαιρία και το θέμα αυτό να αντιμετωπίσουμε, αλλά να προετοιμαστεί σοβαρά και η Κυπριακή Δημοκρατία για το μέλλον. Να μας πει και τι στρατηγική έχει πάνω σε αυτό. Για να μην ξανάρθουμε εδώ μετά από δύο χρόνια και ξανασυζητούμε τέτοια προβλήματα. Και φυσικά να μην απευχόμαστε το να υπάρξουν ατυχήματα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι έτσι επιγραμματικά ανοιχτή παραμένει επιστολή στην, ε, στο Δήμο της Λάρακας, επιστολή στην ε, Κυπριακή Δημοκρατία, τουλάχιστον αυτά. Και από εκεί και πέρα είμαστε σύμφωνοι εμείς και για την επίσκεψη ε, που στο βαθμό που αποφασίσει η Επιτροπή μας, γιατί όχι να δούμε και το θέμα αυτό με μια επιτόπου επίσκεψη. Άλλωστε, όπως συζητήσαμε κύριε Πρόεδρε και το πρωί στους συντονιστές, με βάση και τις διαδικασίες που υπάρχουν, Ήδη συζητήθηκε η αναφορά εν προκειμένου και άρα νομοποιούμαστε αν θέλουμε να κάνουμε και μία επίσκεψη επί του θέματος αυτού για να το διερευνήσουμε στην Κύπρο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Εύη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ συμφωνώ με τους συναδέλφους που θέλουν να μην ανοιχτεί αυτή η αναφορά, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχάς, είμαστε ενώπιον της νιωστής βιομηχανικής εγκατάστασης για την ε, εξόριξη υδρογονανθράκων Θα πρέπει να κατασκευαστούν όλα αυτά με τρόπο ώστε πραγματικά να αλλάξει όψη η Ευρώπη. Και εδώ δυστυχώς τα λόγια μένουν κενά περιεχομένου, ωραία όνειρα, αλλά έπειτα στην πραγματικότητα τα πράγματα διαφέρουν πολύ. Πρέπει να προχωρήσουμε με συγκεκριμένα βήματα στην κατεύθυνση της, απα... της ε, των ρηκτών καυσίμων υπέρ των ανανεώσιμων. Έπειτα δεν είναι αλήθεια ότι πρόκειται για τεράστιες ευκαιρίες απασχόλησης. Και θέλω να αναφερθώ και στην εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας. Μια εφαρμογή που συχνά είναι δυσχερής και ελλειπής. Πέρα από το γεγονός ότι υπάρχουν ε, πάνω άλλες μεγαλύτερες και άλλες μικρότερες εγκαταστάσεις που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογή της οδηγίας ΒΕΖΟ. Αναφέρομαι ας πούμε σε μια κατάσταση που γνωρίζω καλά στη δική μου περιοχή, στη Λομβαρδία, όπου πολλές εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου είτε λειτουργούν είτε κατασκευάζονται και ήδη ευρύνονται καλύπτονται από την οδηγία σε βέζο αυτού του είδους εγκαταστάσεις, ωστόσο δεν υπάρχουν συγκεκριμένα ε, σχέδια για επίγουσες ε, καταστάσεις που είναι απαραίτητες για την προστασία του πληθυσμού. Ο πληθυσμός πολύ συχνά δεν ε, συμμετέχει σε διαβούλευση πριν από την κατασκευή αυτών των εγκαταστάσεων. Δυστυχώς αυτό το γνωρίζουμε και οι κίνδυνοι που μπορεί να αντιμετωπίσουν αυτοί οι πληθυσμοί είναι τεράστια, γιατί εδώ μιλάμε και για σεισμούς, υπάρχουν κίνδυνοι σεισμού, η περιοχή είναι σεισμική. Όχι ότι προκαλούνται σεισμικές δονήσεις λόγω της δραστηριότητας. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν σε θέματα περιβάλλοντος και επιπλέον θα έπρεπε να ακολουθήσουμε το δρόμο της εγκατάλειψης των ορυκτών καυσίμων υπέρ των ανανεώσιμων. Θέλω λοιπόν και εγώ να πω ότι αυτή η αναφορά θα πρέπει να μείνει ανοιχτή, να στείλουμε επιστολή στις τοπικές αρχές, ώστε να τους διαβιβάσουμε τους προγραμματισμούς των αναφερομένων και γιατί όχι στο μέλλον να κάνουμε και μια επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας ώστε να δούμε επιτόπου τι ακριβώς συμβαίνει. Ευχαριστώ. Η κυρία Μολίνα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ την αναφέρουσα για τα όσα μας είπε. Τώρα, έχοντας ακούσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ξέρω, πρόκειται για μία οδηγία ελέγχου. Έτσι όσον αφορά τις επικίνδυνες ουσίες, χημικές ουσίες, πρόκειται για ένα βιομηχανικό λιμάνι 800 μέτρα από πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και φυσικού αερίου και 150 μέτρα από, τις, από τα σπίτια δεν είναι μόνο το περιβάλλον, μα είναι και η ζωή των ανθρώπων που πρέπει να μπουν πριν από οποιαδήποτε άλλη προτεραιότητα ή άλλα άλοθη. Υπάρχει κίνδυνος ή δεν υπάρχει. Μπορεί να υπάρξει σοβαρό ατύχημα, ναι ή όχι. Αυτό είναι που πρέπει να εκτιμήσουμε. Και να αφήσουμε τη γραφειοκρατία και τα άλοθη που χρησιμοποιούμε συχνά. Η σύμβαση του Άρχους για την πρόσβαση στην ενημέρωση από πλευρά των γειτόνων εδώ, σύμφωνα με του ε, γείτονε, δεν ενημερώθηκαν για τη διαδικασία. Καταγγέλουν ότι δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία τη δημόσια διαβούλευση. Γι' αυτό πιστεύω, έχοντα ακούσει του αναφέροντε, ποτέ δεν απευθύνθηκε σε αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεπώ, οι πληροφορίε είναι πληροφορίε τη κυβέρνηση. Όταν λοιπόν θα κρυθεί ένα θέμα και θα γίνει μια έκθεση, θα πρέπει αν μη τι άλλο να έχει μιλήσει κανεί και με τι δύο πλευρέ, όχι με μία μόνο όχι μόνο με τη μία. Δεν είναι αυτός τρόπος να κάνουμε τα πράγματα. Και έπειτα, παρακαλώ, ναι, επιστολή στις Κυπριακές Αρχές, να παραμείνει ανοιχτή αναφορά και να δούμε αν τέλος πάντων θα μπορέσουμε να συμπεριφερθούμε πιο ανθρώπινα, να βάλουμε πρώτα τις ανθρώπινες ζωές και το περιβάλλον και μετά τις επιχειρήσεις, τα οικονομικά συμφέροντα κτλ. Η προτεραιότητά μας πρέπει να είναι σαφής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε παρακαλώ, κύριος Γιάρ. Πρώτη παρατήρηση. Και εγώ συμφωνώ να μην ανοιχτεί η αναφορά. Δεύτερη προκατακτική παρατήρηση. Ήδη από την αρχή του απογεύματος είπαμε ότι δεν θα υπάρξει ούτε ένα μεγάλο έργο που να μην προκαλεί διάσταση απόψεων. Το αν το έργο τώρα οικονομικά είναι αποδοτικό ή όχι, άλλοι λαμβάνουν την απόφαση αυτή, όχι εμείς. Η δική μας ερώτηση είναι οι αρνητικές ενδεχόμενα επιπτώσεις στο περιβάλλον ή στους ανθρώπους. Η Κομισιόν καλά εξήγησε την κατάσταση. Κάπου δεν βλέπω τον διάλογο επιτόπου, την διαβούλευση. Οι δημοκρατικές κοινωνίες όταν υπάρχει ένα πρόβλημα αντιδρούν με διαφάνεια. Δεν θέλουμε να μιμηθούμε τον Πούτιν. Σε αυστηρά διοικούμενες κοινωνίες τα πράγματα πάνε πολύ γρήγορα. Εμείς όμως εδώ χρειαζόμαστε ανοιχτές κοινωνίες, διαφάνεια. Εγώ θα έλεγα λοιπόν να αφήσουμε το θέμα ανοιχτό, την αναφορά ανοιχτή δηλαδή, να στείλουμε μια επιστολή και να πούμε ότι πρέπει να γίνει η διαβούλευση. Εγώ δεν μπορώ να προκαταλάβω οποιαδήποτε έκβαση. Θα πρέπει να γίνει ένα screening, να διευκρινιστεί εάν περιλήφθηκαν ή αν θα περιληφθούν οι τοπικές αρχές και το κοινό. Λοιπόν, να απευθύνουμε μια φιλική αλλά συγκεκριμένη επιστολή στις ε, ε, κυπριακές αρχές και να ζητήσουμε αυτά τα πράγματα και να επανέλθουμε. Έτσι το βλέπω εγώ. Αυτό θα συμπλήρωνα δηλαδή στα όσα, στα όσα είπαν οι συναδελφοί μου. Παραμένει ανοιχτή η αναφορά και παρακαλούμε να αρχίσει διάλογος και να τεθούν τα γεγονότα επί τάπητος. Αυτό όσο μπορώ να κρίνω. Η κυρία Σακοράφα, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. διάβασα με ιδιαίτερη προσοχή και τις 10 αναφορές μπορώ να πω και ε, σε αυτές τις αναφορές αυτό που μπορώ να διαπιστώσω και να επισημάνω είναι ότι γίνονται πραγματικά πολύ σοβαρές και πολύ συγκεκριμένες καταγγελίες από τους αναφέροντες κύριε Πρόεδρε. Ε, ότι δηλαδή το λιμάνι της Λάρνακας μετατρέπεται σε βαρύ βιομηχανικό λιμάνι και γίνονται εργασίες στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αναζήτηση πετρελαίου όπως είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι και φυσικού αερίου. Νομίζω ότι οι κάτοικοι, κύριε Πρόεδρε, δικαιολογημένα διαμαρτύρονται γιατί πρόκειται για την υγεία τους, πρόκειται για την ασφάλειά τους και ακριβώς ε, πρόκειται για, το γεγονός ότι καταστρέφεται μια περιοχή η οποία είναι ε, απείρου φυσικού κάλου και η οποία αποφέρει εκτός των άλλων και ε, οικονομικά ωφέλη όσον αφορά στο τουριστικό επίπεδο. Η αποθήκευση των χημικών ουσιών, όπω λένε στι αναφορέ, η μεταφορά των διενεργών μετάλλων και των επικίνδυνων εκρηκτικών στι πλατφόρμε, ο κίνδυνο τη ρήπανση του εδάφου που θα πρέπει να ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά υπόψη, τη ατμόσφαιρα, τη θάλασσα, πιθανέ διαρροέ χημικών ουσιών και διαδιενέργεια είναι μόνο μερικέ από τι ανησυχίε που αναφέρονται μέσα στι ε, αναφορέ που κάνουν. Στη δε απόφαση του δικαστηρίου, και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε, κύριε Πρόεδρε, όπω αναφέρεται στην περίληψη, επιβάλλεται στι δημόσιε ε, αρχέ όπως χαρακτηριστικά λέει, να λαμβάνουν υπόψη παρατηρήσεις που διατυπώνει το ενδιαφερόμενο ε, κοινό πριν τη λήψη μιας απόφασης και να επεξηγούν τον τρόπο με τον οποίο οι παρατηρήσεις συνεκτιμήθηκαν στην εν λόγω απόφαση. Είναι φανερό λοιπόν πέρα από κάθε αμφιβολία ότι αυτή η διαδικασία δεν ακολουθήθηκε ώστε οι κάτοικοι να γνωρίζουν ποιε συνεκτιμήσει έχουν γίνει για να εκδοθούν οι αποφάσει πολεοδομικών αδειών. Στην απάντησή της η Κομισιόν αναφέρει ότι έχει γίνει διαβούλευση με τους κατοίκους, ενώ αντίθετα οι κάτοικοι ρητά δηλώνουν ότι τέτοια διαβούλευση δεν έχει γίνει προκειμένου να αγκαιωθούν οι άδειε. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, η Επιτροπή μας θα πρέπει να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα που της δίνεται, ώστε να διαπιστωθεί αν έχουν γίνει παραβάσεις οδηγιών, όπως μας αναφέρθηκε προηγουμένως και από την αναφέρουσα, αλλά και από τους συναδέλφους. Προτείνω, λοιπόν, οι αναφορές να παραμείνουν ανοιχτές, να ζητήσουμε με επιστολή μα από τις Εθνικές Αρχές να μας ενημερώσουν πότε έγινε η διαβούλευση και αν υπάρχουν πρακτικά για να μας διαφετούσουν για το θέμα και ποιες περιβαλλοντικές μελέτες υπάρχουν που καθιστούν τις ανησυχίες των πολιτών αβάσιμες, μελέτες τις οποίες, οι οποίες προβλέπονται από τις οδηγίες. Λοιπόν, ε, και τέλος θα ήθελα να, να πω ότι θα πρέπει οι αναφέροντες να μας ενημερώνουν συνεχώς πάνω στα συγκεκριμένα θέματα για να έχουμε συνεχή πληροφόρηση από τη δική του την πλευρά και θα ήθελα επίσης να πω ότι κλείνοντας ότι συμφωνώ και εγώ απόλυτα με το να δημιουργηθεί μια ομάδα ώστε να κάνουμε μια επίσκεψη επιτόπου για να έχουμε ιδία γνώση της κατάστασης η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, σύντομα, να έχετε το λόγο. Ήθελα να κάνω. Ε, δεν υπήρχε δημόσια διαβούλευση. Μια δημόσια διαβούλευση είναι ότι ανταλλάσσονται απόψεις. Εμείς ως κάτοικοι καλεστήκαμε για να μας δώσουν, να μας πούν δεδομένα να μας φέρουν ως δεδομένο την εγκατάσταση των εταιριών στο λιμάνι μας. Αυτό δεν θεωρείται δημόσια διαβούλευση. Ε, δεν έχουμε πάρει μέρος, ε, δεν έχουμε δώσει τις απόψεις μας. Μας το είχαν φέρει δεδομένο αυτό και μας κάνουν το, λιμάνι μας βιομηχανικό χωρίς την δική μας συγκατάθεση ως κάτοικοι της Λάρνακας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, μπορούμε να συμφωνήσουμε το εξή νομίζω. Αφήνουμε ανοιχτή την αναφορά. Και θα στείλουμε τρεις επιστολές. Θέλετε να πάρετε το λόγο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, α, παρακαλώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Ήθελα να πάρω το λόγο για να διευκρινίσω κάποια σημεία τα οποία ανέφεραν ή για να σας δώσω κάποιες επεξηγήσεις αν αυτά που είπα πριν δεν ήταν ξεκάθαρα. Πρώτα απ' όλα, για το ποια οδηγία εφαρμόζεται. Έπρεπε να το είχα αναφέρει. Πάντως και οι δύο οδηγίες έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας. Δεν αλλάζει, είναι διαδικαστικό. Δεν σημαίνει ότι η παλιότερη οδηγία δεν προβλέπει μέτρα για το σχεδιασμό χρήσης γης. Η διατύπωση είναι παρόμοια και το επίπεδο προστασίας είναι το ίδιο. Όσον αφορά την δημόσια διαβούλευση, είπα ότι υπήρξε δημόσια ενημέρωση και σύμφωνα με την ανάλυση μας η οδηγία που εφαρμόζεται εδώ είναι εκείνη για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Και επειδή πρόκειται εδώ για το παράρτημα 2 της οδηγίας, δεν υπάρχει απέτηση βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για δημόσια διαβούλευση. Αλλά οι αρχές οφείλουν να ενημερώσουν τον κόσμο για την απόφασή τους. Οπότε, έγινε αυτό, ενημερώθηκε ο κόσμος. Ένα άλλο σημείο με ρωτήσατε από πού έχουμε τις πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή που βρήκε τις πληροφορίες. Έρχονται από τις προσφυγές που έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμπίπτουν με τόσα λένε οι αναφέροντες. Οπότε αυτά που ακούσαμε από τους αναφέροντες, αυτές είναι, αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε κι εμείς. Μεταξύ άλλων υπάρχει η ανάλυση και του Εθνικού Συνήγορου του Πολίτη, του Κυπριακού. Πρέπει επίσης να επαναλάβω ότι οι πληροφορίες που πήραμε δεν καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει παραβίαση του περιβαλλοντικού νόμου. Και ένας αξιότιμος ευρωβουλευτές είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι υπήρχε παραβίαση. Όχι, εμείς δεν έχουμε εντοπίσει παραβίαση. Δεν είπε ότι υπάρχει παραβίαση. Δεν έχει εντοπιστεί. Από εκεί και πέρα θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά την οδηγία σε βέζο. Τι συμβαίνει εδώ. Αυτές οι καταστάσεις δεν εμπίπτουν στα πλαίσια της οδηγίας σε βέζο, δεδομένου του μέγεθος και των πληροφοριών που έχουμε σχετικά. Το μόνο θέμα που έπρεπε να εξετάσουμε ήταν το κατά πόσο τίθεται ζήτημα με τις άλλες τις παλιότερες ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις που βρίσκονται εκεί κοντά στο λιμάνι της Λάρνακας. Και είναι οι εθνικές αρχές αυτές οι οποίες πρέπει να διασφαλίσουν ότι υπάρχει αρκετή απόσταση από αυτές. Δεν έχουμε πάρει καμία πληροφορία σύμφωνα με την οποία να μπορούμε να καταλήξουμε στο αντίθετο συμπέρασμα, ότι δηλαδή οι εθνικές αρχές δεν έχουν φροντίσει να υπάρχει η απόσταση αυτή. Ελπίζω έτσι να ξεκαθάρισα τα πράγματα. Και αν έχετε κάποια άλλη απορία, τότε ευχαρίστω να σας δώσω και άλλες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο για όλους ότι δεν μπορούμε να την κλείσουμε αυτή την αναφορά σήμερα. Συμφωνούμε λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή. Συμφωνεί. Και συμφωνούμε και για τις τρεις επιστολές που είπαμε ότι θα γράψουμε. Θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει γραπτά λεπτομέρειες για την απόψη της όσον αφορά αυτό το θέμα. Άλλη η επιστολή είναι να ζητήσουμε από το Υπουργείο της Κύπρου να μας ενημερώσει επίσης και η τρίτη επιστολή θα είναι προς το Δήμο για να ζητήσουμε και εκεί πληροφορίες από το Δήμο να δούμε τι μας λέει. Σημειώνουμε επίσης και τη δυνατότητα να υπάρξει κάποια αποστολή μελέτης. Εκεί δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε τώρα, οι συντονιστές εννοείται θα το συζητήσουν αυτό. Ωραία. Κυρίε και κύριοι, συνεχίζει στα αγγλικά ο πρόεδρο. Τίποτα άλλο. Σα ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σα ε, εδώ και ιδιαίτερα ευχαριστώ για τη διερμηνία, λέει ο Πρόεδρο. Καλό βράδυ σε όλους. Και κλείνουμε τη συνεδρίασή μας για σήμερα το βράδυ.